Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι δεν είναι πολλά τα μέλη εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αγαπητέ φίλε, σας ευχαριστώ που ήρθατε η κυρία Σάντριν μόνη από ό,τι βλέπαμε και εγώ. Α, κι άλλο ένα μέλος. Δύο λοιπόν και εγώ τρεις. Πολύ ωραία. Α, είστε κι εσείς, ναι, συγγνώμη. Τέσσερις. Είναι τελικά αρκετοί οι συνάδελφοι. είναι και ο εισηγητής μας, ο κύριος Γιάβορ. Λοιπόν, σημείο 1. Θα θέλαμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια μπορούμε να την εγκρίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σας κάνω σε πέρα ανακοινώσεων του Προέδρου. Να εγκρίνουμε τα πρακτικά 11-12 Ιουλίου και 15 Σεπτεμβρίου 2016. Υπάρχουν σχόλια για τα πρακτικά? Όχι. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. the title, which is very long. Ο τίτλος είναι κάπως μεγάλος. Ένα λεπτό θα κρατήσει και μόνο, μόνο τίτλος. Λοιπόν, για τις μειώσεις, μειώσεις των εκπομπών αγριών του θερμοκηπίου από τα κράτη-μέλη από το 2021 στο 2030 για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και τροποποίηση του κανονισμού υπαρθμών 525 κάθετος 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Αγαπητέ Μπένεντικτ, ο τίτλος είναι τόσο μεγάλος που πρόλαβες να φτάσεις εδώ στην Επιτροπή μας τον Οκτώβριο του 2014 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισαν ε, έναν στόχο δεσμευτικό για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 40% μείωση και κάποιοι τομείς ε, δεν καλύπτονται από το ETS, πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 30% έως το 2020, σε σχέση με το 2005 πάντα, για να συνεισφέρουν τον συνολικό στόχο. Ο προτινόμενος κανονισμός μεταφράζει αυτήν τη δέσμευση σε συγκεκριμένους δεσμευτικούς στόχους για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2021-2030. Με τις αρχές της ε, περιολικής ακαιρεότητας, της σωστής σχέσης της κόστης ωφέλους και της ε, δίκαιης κατανομής και βεβαίως ε, η υπεύθυνη επιτροπή είναι η Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ο συνάδελφος, ο κύριος Γκερμπράντη της Άλντε είναι ο εισηγητής. Είναι και ένα πληρωματικό μέλος της Επιτροπής μας. Οπότε ο βασικός εισηγητής ο δικός μας είναι από την Επιτροπή Ήτρε ας πάμε στη δική μας συζήτηση. Θα πάμε στη συζήτησή μας τώρα. Θα ήθελα ο εισηγητής μας, ο Μπένεντικτ Γιάβορ, από την Γκούε, να μας παρουσιάσει την άποψή του. Ευχαριστώ πρόεδρε, εξωπροσπώ τους πράσινους ε, και όχι την ΚΟΕ. Βεβαίως, ε, πόσο είναι κλιματικό ζητήμα το πράσινος θα ήσασταν και γκου να ήσασταν δεν έχει σημασία, λέει ο κύριος Γιάβορ, ποιο κόμμα εκπροσωπώ, η δουλειά με τους κοιόδους συγκητέ ε, θα προχωρήσει με βάση αυτή την προσέγγιση. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Κατάφερα τελικά να έρθω και έχω ένα δύσκολο απόγευμα και σε άλλες επιτροπές παραλλήλως. Όπως περιγράψατε πολύ σωστά, η Επιτροπή Ήτρε εδώ θα δώσει μια γνώμη προς την Επιτροπή Ένβη που είναι η ε, βασική Επιτροπή για το θέμα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα που είναι σημαντικά για την Επιτροπή Ήτρε ιδιαίτερα και τα μέλη της να τα τονίσουμε δηλαδή και να συνεισφέρουμε στο μέτρο του δυνατού για να φτάσουμε σε έναν όσο γίνεται καλύτερο κανονισμό σε συνεργασία με την Επιτροπή Ένβια αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της προσπάθησε να λάβει υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού και τις ε, εξελίξεις που απορρέουν από εκεί, τις επίγουσες δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού Ναι, μάλλον θα πρέπει να αλλάξουμε, λέει ο πρόεδρος, τη σειρά στα κανάλια. Στο 2 θα πρέπει να είναι τα αγγλικά. a different language. But you can, you can speak because the native language is also channel zero. Please, the floor is yours. If you don't mind, I continue in English, of course. Ναι, συνεχίζω. Μπορώ να μιλήσω για τη μητρική μου βέβαια, αλλά συνεχίζω στα αγγλικά. Είναι πιο εύκολο για όλους νομίζω να παρακολουθούν τα αγγλικά σε σχέση με την όμορφη ουγγρική γλώσσα. Λοιπόν, πρέπει να σεβαστούμε τη Συμφωνία του Παρισιού. Η πρόταση της Κομισιόν έρχεται να απαντήσει σε αυτές τις απαιτήσεις, αλλά μερικώς. Θεωρώ ότι πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε σχέση με το πακέτο για το περιβάλλον ε, και την ενέργεια για να μπορέσουμε να πετύχουμε το τον στόχο των 1,5 βαθμών ε, Κελσίου για την κλιματική αλλαγή όπως ε, τέθηκε αυτό ως στόχο στη Συμφωνία του Παρισιού. Βεβαίως θα φανεί σαφέστερα σε τι είδου συμφωνία μπορούμε να φτάσουμε στου κοινού συζητητέ αργότερα. Αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη συνεργασία μα σε επίπεδο ήτρε. Οι εκπομπέ φαινομένων θερμοκηπίου αναμένεται να μειωθούν από το 2016 στο 2020. Έτσι λοιπόν η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την παρούσα μορφή ενδεχομένω να μα δώσει την ευκαιρία ε, να έχουμε μια αύξηση του ε, προπολογισμού για τον άνθρακα, η οποία δεν χρειάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επαληθεύσουμε, δεν θα, δεν επιβραβεύσουμε χώρες που δεν ε, πληρούν τους στόχους. Θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται στις προσπάθειες ε, του κάθε κράτους μέλους. Εκτιμώ ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οποιαδήποτε βελτίωση σε σχέση με άλλες περιόδους πάνω από το 2020 θα ακυρώνεται. Δεν θα υπάρξει μεταφορά ε, σε ό,τι αφορά τις εκπομπές θερμού αέρα θα υπάρχει μια αύξηση στου τάξεω των 25 δισεκατομμύριων τόνων έω το 2020. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ευελιξία. Αυτό είναι αναγκαίο, έτσι ώστε να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταυτόχρονα δεν πρέπει να δημιουργήσουμε κενά. Ευελιξία ναι, ε, αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος για να βοηθήσει τα κρατημέλη να πετύχουν τους στόχους, αλλά δεν πρέπει να ε, δημιουργήσουμε καταστάσεις όπου τα κράτη-μέλη θα βρίσκουν τρόπους να παρακάμψουν τις υποχρεώσεις τους. Στο σχέδιο γνωμοδότησης θα ζητήσω να υπάρχουν και έλεγχοι ε, πρόορης ε, Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο να υπάρχει ένας κανονισμός, αλλά να υπάρχει μια παρακολούθηση στη συνέχεια κατά την υλοποίηση, κατά την εφαρμογή. Θα πρέπει να ελέγξουμε πώς τα κράτη-μέλη λοιπόν συμμορφώνονται με τον κανονισμό αυτόν. Χρειάζεται ένας ε, ισχυρός μηχανισμός ε, αναθεώρησης, επανεξέτασης, ε, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα όπου διαπιστώσουμε κενά. Μόλις το 2027 θα γίνει ο πρώτος έλεγχος συμμόρφωσης, αυτό προτείνει η Κομισιόν, οπότε δεν θα υπάρξει χρόνος για περαιτέρω πολιτικές εφόσον δούμε ότι έχουμε αποκλίνει από το στόχο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ετήσιους ελέγχους συμμόρφωσης όπως υπάρχουν και ετήσιες ε, εκθέσεις για τις εκπομπές αλλά και διετής εκθέσεις για τις προβολές ε, δεν δημιουργεί αυτό περαιτέρω διοικητικό άχθο. Εν πάση και αν το δημιουργεί, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί πρέπει να έχουμε τέτοιου ελέγχου Κάτι άλλο που θα συζητήσουμε και ως συγητές κατά τη διάρκεια των ε, επαφών μας. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα μάλλον, αλλά αυτές είναι οι πιο βασικές προκλήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να έχουμε ένα κανονισμό που να είναι φιλόδοξος, που να μοιράζει σωστά την προσπάθεια να πετύχουμε να σεβαστούμε τις απαιτήσει των συμφωνίας του Παρισιού, να έχουμε και κατά νου βεβαίως και τις αρκετά ε, σοκαριστικές εξελίξεις ε, στην στον Αρκτικό ωκεανό ε, που αποδεικνύουν ότι πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε ένα όσο γίνεται πιο φιλόδοξο κανονισμό για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Αν δεν το πράξουμε αυτό, είναι πιθανό το συνολικό παγκόσμιο ε, κλιματικό σύστημα να καταρρεύσει. Από κοινού με του και όλου λοιπόν, ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ήτρε που να βοηθάει την Επιτροπή Ένβη να επηρεάσει την πρόταση της Κομισιόν προς μια κατεύθυνση που να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να έχουμε ένα κανονισμό που να οδηγήσει μια πραγματική κατανομή της προσπάθειας ε, για να μπορέσουμε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Σα έδωσα λίγο παραπάνω χρόνο. Και τώρα... Η κυρία Κομπούλα Νάτσι. Ευχαριστώ. Έχετε τα χαιρετίσματα τη Σιμώνα που έχει κολλήσει στην Ιταλία στο αεροδρόμιο. Ε, αυτός ε, ο κανονισμός αποτελεί άλλη μια ε, σημαντική νομοθεσία μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Εμείς στην Ήτρε θα το συζητήσουμε, θα συζητήσουμε τις συμβολές των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για την εξάλληψη της χρήσης του άνθρακα σιγά σιγά. Μιλάμε για μεταφορές, κτίρια, γεωργία αλλά και διαχείριση αποβλήτων. Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει στο να υπάρξει μείωση 30% των ευρωπαϊκών εκπομπών σε σχέση με το επίπεδο του 2005. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος που συνδυάζει την ε, βιομηχανική μετατροπή με ε, την χρήση ανανεώσιμων πηγών. Υπάρχουν εντυπωσιακέ επιπτώσει των κλιματικών αλλαγών, αυξάνεται ο διεθνή ανταγωνισμός για λοιπεί πόρου και γι' αυτό και δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να περάσει. Α σκεφτούμε αυτέ τι τεχνολογικέ εξελίξει στον τομέα των μεταφορών και στην παροχή καυσίμων, τα νέα σύνορα για τα νέα κτίρια και τέλο, να μην ξεχνάμε και την ε, πρόοδο του ε, σχεδιασμού στα προϊόντα για τα εισπρότεση ύλες για την επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο θα πρέπει να διευκολύνεται ε, αυτή η προσπάθεια με ένα μακρόπνο ε, σχέδιο, νομοθετικό πρόγραμμα, το πλαίσιο, η, απόφαση πλαίσιο για την κυκλική οικονομία, ε, το ETS κτλ, καθώς και τις προτάσεις που θα προέλθουν από την Κομισιόν μέσα στο νέο χειμερινό πακέτο. Σε σχέση με αυτά μπορούμε να συμβάλλουμε στο Κοινοβούλιο προσθέτοντας την αλληλεγγύη και τη συνοχή στις προτάσεις της Κομισιόν. Δύο σημαντικές πτυχέ θέλω λοιπόν να τονίσω. Πρώτα, η πρόταση της Κομισιόν είναι αρκετά φιλόδοξη δεδομένου του νέου μηχανισμού ευελιξίας, όπως ε, ανέφερε και ο εισηγητής μας ε, Γιάμπορα. Θα πρέπει να αναλάσουμε το δυνητικό αντίκτυπο αυτών των νέων ευελιξιών που συνδέουν το ETS με την ε, γενικότερη προσπάθεια και το project για τη μείωση μέχρι το 2050, καθώς και τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβάλουμε μετά από τη Συμφωνία του Παρισιού. Άλλο σημαντικός ε, παράγοντας είναι η ειδική κατανομή. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη δικαιωτική κατανομή για αυτές τις προτάσεις. Έχουμε δύο σημεία σημαντικά. Το ένα είναι ο μηχανισμός ευελιξίας, που ασυμμετρικά κατανέμει στα κρατημέλη και δεύτερον, οι στόχοι από το, συγκεκριμένοι από το 2020 και μετά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά των κρατών μελών, να υπάρξει ισορροπία ώστε να οθηθούν, να παροτριθούν τα κράτη μέλη να λάβουν δράση. Σας ευχαριστώ πολύ και εξ ονόματος της Άλντε θα δώσω το λόγο στην κυρία Βουντσέτ. Αφού μελέτησα το κείμενο, να πω ότι η πρόταση της Κομισιόν για τη μείωση των εκπομπών ε, στους λόγω τομείς είναι καλό αρχικό κείμενο, ωστόσο πρέπει οπωσδήποτε ε, το Ευρωκοινοβούλιο να προσθέσει περισσότερη φιλοδοξία στο κείμενο. Θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μείωσης των εκπομπών όπως αυτοί ε, συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο του Παρισιού. Σε αυτό το έγγραφο περιλαμβάνονται επίμαχα ζητήματα που όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να τα βελτιώσουμε, αλλά δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για διαπραγμάτευση διαπραγμάτευση. Ένα παράδειγμα είναι τα ποσοστά που αναφέρονται στη μείωση εκπομπών για κάθε χώρα. Υπάρχουν δύσκολες ισορροπίες εκεί ε, επίσης είναι αλήθεια ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να, βελτιωθούν, να βελτιωθεί η κατάσταση, όμως δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για διαπραγμάτευση και επίσης πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο, όσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο μάλλον για διαπραγμάτευση, τόσο καλύτερο. Και το μέσο της γεωργίας είναι ένας από αυτούς ότι πρέπει να γίνει ε, διαπραγμάτευση. Δεν θα πρέπει να μείνει η γεωργία στο περιθώριο της ενεργειακής ε, μετάβασης. Ε, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το ρόλο της Γεωργίας όσον αφορά την μείωση των εκπομπών και την συγκράτηση των ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να συμβάλλει στη μείωση, αλλά να σκεφτούμε ότι και στο μέλλον αν δεν κάνουμε κάτι οι εκπομπές από τον τομέα της Γεωργίας θα αυξηθούν. Θα πρέπει λοιπόν η Γεωργία να συμβάλλει ενεργά στην μείωση. Και εξάλλου το μέσο τη Γεωργία μπορεί να το καταφέρει αυτό παραμένοντα ανταγωνιστικό και αποδοτικό. Δηλαδή αντικαθιστώντα, α πούμε, την συμβατική γεωργία από την βιολογική. Που σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ε, λιπασμάτων και ε, ζυζανιοκτώνων. Επίση σημαντικό είναι το θέμα τη ευελιξία στην πρόταση της Κομισιόν που επιτρέπει αντιστάθμιση των εκπομπών σε ανταλλαγή με την αναδάσωση. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια καλή ιδέα, μπορεί όμως να καταλήξει ανεπαρκές ο σύστημα γιατί η κοπή, η αποψήλωση δασών μπορεί τελικά να ξεπεράσουν ε, την αναδάσωση που μπορεί να δίνει δικαίωμα σε αντιστάθμιση. Να υπάρχουν δηλαδή σαφή κριτήρια στην πρόταση που θα προστατεύουν την ε, χρήσιμη, το χρήσιμο βίο αυτών των νέων δασών. Αν δεν υπάρχουν εγγυήσει για αυτές τις δασικές εκτάσεις ότι θα ζήσουν ας πούμε, για τα δε χρόνια, ε, υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθούν. Ε, οι διατάξεις αυτές. Και έπειτα, προθεσμία για αναθεώρηση. Το πρόβλημα είναι ότι η αύξηση τη προθεσμία είναι υπερβολική, γιατί αντί να γίνεται αναθεώρηση κάθε χρόνο, εξέταση μάλλον κάθε χρόνο, λέει να γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Αυτό είναι υπερβολικό. Η στόχη η αιτήση, θα πρέπει να αιτήσει, γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε περιθώριο να αντιδράσουμε αν τα κράτη-μέλη ε, αποκλίνουν. Γι' αυτό νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνεται ένα έλεγχο τουλάχιστον κάθε δύο ή τρία το πολύ χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφο Μπένσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Σονκέλη δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Και θέλει να σημειώσει ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει τον έλεγχο αυτής της προσπάθειας η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τηρηθούν οι συμφωνίες των Παρισίων και να αναλυφθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες για την πολιτική με την εξορρόπηση των δεσμεύσεων για τη συγκράτηση των κλιματικών αλλαγών και, των, ε, και πάντα με προστασία των ιδιαιτεροτήτων των, ε, των οικονομιών μας ε, που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση κίνησης. Η πρόταση λοιπόν συνιστά μια ισορροπημένη πρόταση, φιλόδοξη. Και είναι σημαντικό η ευελιξία αλλά και κίνητρα για πραγματικές δράσεις να υποστηριχθεί. Ευελιξία λοιπόν για τα κράτη-μέλη μαζί με τις προτάσεις για νέες ευελιξίες με το Λούλου CF ε, ε, ε, και τις πιστώσεις των εκπομπών. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν μεγάλο μερίδιο στις εκπομπές από τη γεωργία. Έχουμε λοιπόν την ιδέα της βιώσιμης διαχείρισης γης, της προστασίας από την αποψηλού των δασών, και μέτρα για τη συγκράτηση του άνθρακα. Τα κράτη τα οποία έχουν ήδη ε, αναπτύξει σημαντικά προγράμματα για την προστασία των δασών τους πρέπει να στηριχθούν. Πρέπει να αποτραπούν επίσης ε, εκείνες οι δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις εκπομπές. Το ETS και οι λοιπές δράσεις εκτός ETS πρέπει να συνδυαστούν για τον ίδιο στόχο. 40% μείωση των ακουμπών στο 2030. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για πλήρης πιστώσεις ETS επιτρέπει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα το οποίο σημαίνει και στήριξη των κρατών μελών στις ε, προκλήσεις που έχουν μπροστά τους ορισμένα κράτη ενώπιον του 2030 και εν γέννη αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη βελτίωση της πρότασης με ουσιαστικές μειώσεις εκπομπών στους τομείς εκτός ETS. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Διευθυντής εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης για τις Κλιματικές Αλλαγές, ο κ. Μέτσικερς, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Είχαν όλοι πιστεύω το χρόνο να εξετάσουν την πρόταση. Και βεβαίως ευχαριστούμε τους βουλευτές που κρίνουν ισορροπημένοι και ε, ως προς το περιβάλλον και ως προς το κόστος την πρόταση. Ορισμένες μόνο παρατηρήσεις για τα επιμέρους σημεία. Θα ήθελα ξεκινώντας να καθησυχάσω τον προηγούμενο μιλητή σε σχέση με τις ε, υπερβολικά υψηλές επιδόσεις προηγουμένου, της προηγουμένης περίοδου δεν πρόκειται να μεταφερθούν. Δεν προβλεπόταν τους άλλους, δεν ζητούμε τροποποίηση. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης δεν πιστεύουμε ότι κάποιο κράτος μέλος κινδυνεύει να μην τηρήσει τους στόχους του για το 2020. Αυτό θα έχει μεγάλο κόστος. Υπάρχει ένας βαρύς μηχανισμός προσαρμογής ε, στις διατάξεις αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσει να ισχύει. Ε, νομίζω ότι σε σχέση με τις επικρίσεις ότι είναι περίπλοκο το σύστημα δεν επιτρέπει παραθυράκια ή κενά στην νομοθεσία. Είχε μια συνεπίσταση στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κείμενο συμμόρφωσης. Θέλουμε, πιστεύω, να προχωρήσουμε προς ένα ε, ευθυγραμμισμένο, ένα εξομαλυμένο ε, σύστημα το οποίο δεν θα φέρνει τα κράτη-μέλη ενώπιον της σχολιών, άρα έχουμε μέτρα τόσο ήπιας όσο και αναγκαστικής νομοθεσίας. Τα ήπια μέτρα είναι ότι κάθε χρόνο θα ε, επαληθεύουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να τηρήσουν τι δεσμεύσει τους, αλλά δεν θα τα ε, προσάγουμε στο δικαστήριο κάθε χρόνο σε περίπτωση μη τηρήση των δεσμεύσεων. Θα του υπενθυμίζουμε πάντως την θέση στην οποία βρίσκονται σε σχέση με την Ενεργειακή Ένωση και ενδέχεται μια φορά στα πέντε χρόνια με το σύστημα της σκληρής επιβολής των μέτρων της αναγκαστικής δηλαδή νομοθεσίας να τα παραπέμπουμε σε δίκη εάν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Επίσης, ύστερα από μια πενταετή χρονική περίοδο μπορούμε να εξετάσουμε την πορεία του ETS και άρα να προσαρμόσουμε γιατί σε αιτήσια βάση δεν είναι δυνατόν να γίνεται ε, συμμόρφωση και αναπροσαρμογή στον τομέα της γεωργίας ειδικά. Για την ε, Ελαφριά υλοτόμηση, παρανόμη υλοτόμηση, αυτό δεν καλύπτεται τη συγκεκριμένη πρόταση. Υπάρχει άλλη πρόταση που θα σας απασχολήσει μετά τις 5 από ό,τι βλέπω σήμερα και με την οποία στόχος είναι, εάν γίνεται υλοτόμηση, να καταγράφεται και αυτή στο ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά νομίζω. Α, όχι, υπήρχε ακόμη ένα σχόλιο ότι ε, η γεωργία απαλλάσσεται κάθε ευθύνη. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Η γεωργία θα πρέπει να συνεχίσει να περιορίζει τις εκπομπές της μέσω και του συστήματος επιμερισμού της προσπάθειας. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί. Ωστόσο θέλουμε και στους γεωργούς να δώσουμε τη δυνατότητα να εξετάσουν τις δυνατότητες που έχουν ε, για περιορισμό των εκπομπών τους στον τομέα LULUCF. Και άρα είτε με το ε, ένα σύστημα είτε με το LULUCF θα έχουμε αυτή την ε, ιδέα μιας γέφυρας που θα τους επιτρέπει να περιορίζουν τις εκπομπές. Δεν θα μείνει όμως κανένας τομέας ε, άμυρος ευθυνών ή απαλλαγμένος από την υποχρέωση τήρησης. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τα σχόλια. Για το τέλος της συζήτησης, αν θέλει ο εισηγητής μας, Έχετε 7,5 λεπτά χρησιμοποίηση στην εισαγωγική σας παρατήρηση. Αν θέλετε το πολύ 30 για τα 7,5 λεπτά στην ομάδα μας, στην επιτροπή μας είναι ρεκόρ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και τους για τις συνεισφορές τους, αλλά και τις εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ε, προφανώς ε, θα συνεργαστούμε με τους συζητητές έτσι ώστε να μπορέσουμε όντως να βελτιώσουμε το κείμενο στην Επιτροπή μας και ελπίζω να σταθεί από επιτυχία το έργο μας. Ναι, ήσασταν πολύ καλός, αλλά να είστε και πιο σύντομος. Να περάσουμε τώρα στο χρονοδιάγραμμα την μέσα διάταξη. Το Μάρτιο θα ψηφιστεί ε, στην Επιτροπή 29 Μαΐου στην Ένβη. Θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα, να είμαστε έτοιμοι δηλαδή τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ψηφοφορία στην Ένβη για να επηρεάσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 5 της διάταξης, σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. Η συγγήτριά μας είναι η, Αγγέλικα Μλίναρ από την Άλντε. Να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση τον Απρίλιο του 2016, πριν από έξι μήνες περίπου, είναι το σχέδιο δράσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. Αυτό το σχέδιο δράσης έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου για την περίοδο 2011-2015 για μία πενταετία λοιπόν η Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι η βασική επιτροπή για την προπαρασκευή της νομοδότησης πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου αλλά στα πλαίσια του κανόνα 54 ε, συμμετέχει η Ήτρε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιες αποκλειστικές αρμοδιότητες για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Και εδώ έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας ε, για το ζήτημα αυτό. Να ζητήσω λοιπόν από την Αγγέλικα να κηρύξει την έναξη των συζητήσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που θα γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό σήμερα και βεβαίω αν, υπομονώ να, συνεργαστώ με του και συγητέ για το θέμα αυτό, όπω είπε ο πρόεδρο, έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για μια σειρά αποζητήματα σχετικά με αυτή την γνωμάτωση πρωτοβουλία. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι βασικό στοιχείο ε, τη ε, στρατηγική για την ψηφιακή αγορά. Μειώνεται το κόστο, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, μειώνεται το διοικητικό άρθρο και για τι επιχειρήσει και για του εργαζόμενου. Ε, πολλά και του φορολογούμενου πολίτε. Ε, πολλά θα μπορούσαν να υποθούν, αλλά θα αναφερθώ στα βασικά. Αναμένω ότι έχουν και του αδέλφους να ακούσουν τι απόψει του. Καλωσορίζω ιδιαίτερα την ανακοίνωση αυτή για το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ανέφερε και ο πρόεδρο. Πολλά έχουν γίνει ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διευκολύνουμε την ψηφιακή μετάβαση τη διακυβέρνηση. Ε, έχουμε τον κανονισμό, έχουμε το e-procurement. Είναι μια σειρά από νομοθετήματα που οδηγούν σε απλοποίηση και για τους πολίτες, αλλά εξασφαλίζουν και το συντονισμό. Η εξολόγηση αντικτύπου και ενδεχόμενη αναθεώρηση της υπάρχους, του υπάρχοντας πλαισίου διαλειτουργικότητας ε, έχουν ξεκινήσει και αυτά είναι καλοδεχούμενα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σαφές, ε, συνεκτικό ε, σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι νέε τεχνολογίε που εξελίσσονται πολύ γρήγορα να λαμβάνονται υπόψη σε ό,τι αφορά το θέμα τη διαλειτουργικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα μέσω του συντονισμού με τα κράτη-μέλη για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό κατάλογο προτύπων ICT για τι δημόσιε προμήθειε. Όμω, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο πλαίσιο για την ε, ψηφιακή ε, μετάβαση της διακυβέρνηση, θα πρέπει να, οι ε, να αντέχουν στο μέλλον πρέπει να είναι, να είναι ανοιχτές ε, προς τον χρήστη, φιλικές προς τον χρήστη μάλλον, να είναι ανοιχτές. Είναι πολύ ε, γρήγορε ε, οι εξελίξει, οι, οι τάσει, το cloud computing. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ανοιχτοί. τα open data μπορούν να μας βοηθήσουν για τη δημιουργία νέων λύσεων, νέων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα Βεβαίω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων και τη ιδιωτική ζωή των συμπολιτών μα. Θα πρέπει επίση να επικαιροποιήσουμε τις υπηρεσίες μέσω των πολιτών ε, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σχετικές υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο φιλική προς το χρήστη και μια προσέγγιση και μια προσέγγιση που να επικεντρώνεται στο χρήστη. Θα πρέπει λοιπόν οι υπηρεσίες να είναι ψηφιακά προσβάσιμες στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η ίδια η ιστοσελίδα και άλλα θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ε, της ε, αλλαγής, της αλλαγής. Το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι καινοτόμο, πρέπει να κοιτάς προς το μέλλον, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να εφαρμοστούν αυτές οι δράσεις. Ε, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε υποδομέ, ε, η ποιότητα, ο ανοιχτό χαρακτήρα, η διαλειτουργικότητα, η ασφάλεια των δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ενισχυμένε ε, υπηρεσίε με τι επιχειρήσει, με του πολίτε, να χρησιμοποιήσουμε τα ανοιχτά δεδομένα διακυβέρνηση και να κάνουμε καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσω τα σχόλια των αδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ, η κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επικοινωνική διοίκηση αποτελεί ένα τεράστιο δυναμικό για την ε, ανανέωση των σχέσεων ανάμεσα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τη μια πλευρά και τις δημόσιες αρχές από την άλλη. Η ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών επιτρέπει σε όλους να κερδίσουν χρόνο, χρήμα, αλλά και αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Αυτό επιτρέπει επίσης να μειωθεί η γραφειοκρατία, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες μας και για τις, ε, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στηρίζω λοιπόν την ε, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο δράσης που ακολουθεί το σωστό δρόμο. Ε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή συνεργασία για να εξασφαλίσουμε την διαλειτουργικότητα πέρα από τα σύνορα. Επίσης, ε, συμφωνώ με τις διάφορες αρχές του σχεδίου, ψηφιακή ε, ε, χρήση, εξορισμού, αδιαλειτουργικότητα, ανοιχτά δεδομένα και κρατικοί διαγωνισμοί επιγραμμικά επίσης. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρχουν και τα απαραίτητα μέσα και θέλω προ αυτό να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι η εμπιστοσύνη είναι το κύριο συστατικό της επιτυχία. Θα πρέπει πραγματικά οι χρήστε και οι εταιρείε να ε, αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις διοικήσεις ε, για την προστασία των ψηφιακών τους δεδομένων. Δεύτερο σημείο που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ψηφιακή ένταξη όλων. Δηλαδή η ηλεκτρονική δικυβέρνηση θα πρέπει να, ξε, 100% την, ε, την ε, παλαιού τύπου διοίκηση, γιατί ας πούμε στις αγροτικές περιοχές ή για τους πιο ηλικιωμένους ή τους ανθρώπους με αναπηρία ή αυτούς που δεν είναι εμπειροί και εξοικειωμένοι, ε, θα πρέπει να υπάρξει και να μην δημιουργηθούν ε, ρήγματα ε, ψηφιακού τύπου. Επίσης, ε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι στην εξυπηρέτηση του χρήστη, δηλαδή να είναι εύχρηστη φιλική προς τον χρήστη. Και τέλος, να πω ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως είπε και η συνάδελφος, θα οφείλουν να δώσουν το παράδειγμα και ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μεταφράζοντας ε, τους ε, ιστοτόπους ε, των ευρωπαϊκών θεσμών στις διάφορες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι σήμερα όλα είναι στα αγγλικά και δεν ε, μιλούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες στην αγγλική. Εάν θέλουμε λοιπόν να είναι προσβάσιμοι οι ιστότοποι, πρέπει να γίνει και εδώ μια παραπάνω προσπάθεια. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Ε, περιμένουμε ονικομονησία το σχέδιο γνωμοδότησης της ε, συναδέλφου Μίλναρ και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Και εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Περνάμε στην ομάδα των σοσιαλιστών και τον συνάδελφο Ζωρίνιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια ως σκιώδης εισηγητής για του σοσιαλιστές να τη πω ότι μπορεί να βασίζεται στην ενεργή μου συνεργασία ε, και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα κάποιες σκέψεις, ε, κάποιου προβληματισμού για αυτό το σχέδιο και την ένταξη, την, το συνδυασμό μάλλον αυτού του σχεδίου με άλλε πρωτοβουλίε για την ψηφιακή ατζέντα. Ξέρουμε ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση και είναι αυτός κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωσή μας. Πρέπει να βασιστούμε στι ανθρωπιστικέ αξίε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα δημοκρατικά δικαιώματα συμμετοχή. Και αυτέ οι αξίε εδώ έχουν μια τεράστια ευκαιρία μέσω τη ε, ψηφιακή διακυβέρνηση. Μπορούμε να φτιάξουμε μια βάση Ευρωπαϊκή ταυτότητα που να μα διαφοροποιεί. Και αυτό η διαδικασία γίνεται με το πρόγραμμα Square, για το οποίο ήμουν εισηγητής και που αφιερώνει ακριβώς ε, την προσπάθειά τους σε δημιουργία κοινών ε, βάσεων, ε, όπου θα μπορούν να ακολουθήσουν τεχνολογική πρόοδο. Τα πράγματα αυτά μετατρέπονται γρήγορα, αλλάζουν γρήγορα. Πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε εμείς αυτές τις, τις, τις διαδικασίες, όπου γρήγορα να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές αυτές και τις καινοτομίες. Επίσης έχουμε το project για την δυνατότητα μεταφοράς και το συζητήσαμε σε αυτήν την Επιτροπή και ε, έχουμε και το Wi-Fi για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο πρόγραμμα για το οποίο είμαι επίσης εισηγητής για τον ίδιο λόγο και είναι εδώ μια πρόκληση που απευθύνω σε όλη την ομάδα που θα εργαστεί για αυτό εδώ το σχέδιο, ότι η αρχή πλήρης δηλαδή ηλεκτρονική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να έχουμε δημόσιες διοικήσεις ε, ανοιχτές για όλους και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους ε, ανθρώπους. Βεβαίως αυτό δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες στις εταιρείε. Πάντως ε, μπορούμε να σηματοδοτήσουμε την ε, διαφορά και να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο ώστε να επιτύχουμε σε αυτή τη νέα φάση της ψηφιακή μας μετάβασης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ συνάδελφε, ο κύριος Ραϊμόν των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η έκθεση και το γενικότερο θέμα μπαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε θετικά με την έκθεση αυτά. Σε τρία σημεία θα ήθελα να σταθώ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχω την εντύπωση πως το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν ήδη πρωτοπόρο ρόλο, έχουν προτείνει τις εντολές. Νομίζω ότι μπορούν να διαμορφωθούν αυτές ακόμη πιο, ε, με τρόπο ακόμη πιο διαφανές. Διαφανή, πάντως πρέπει να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι το γεγονός ότι για τα κράτη-μέλη υπάρχουν εθνικές αρμοδιότητες, διαφορετικά πολλές φορές συστήματα με διαφορετικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις, ακόμη και καταγραφόμενα δεδομένα μπορεί να είναι διαφορετικά από κράτος σε κράτος. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να πιέσουμε ως το δυνατό, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ε, ομοιότητα στα συλλεγόμενα στοιχεία, μακροπρόθεσμα, και βεβαίω, αν θέλουμε να προχωρήσουμε ως Ευρώπη μαζί, θα πρέπει να υπάρχει ένας απλός τρόπος για τον πολίτη να διαβάσει το σύστημα. Και για την τρίτη μου παρατήρηση, Στο ε, σχέδιο της Επιτροπής βλέπουμε ότι η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις. Ναι, βεβαίω δεν το αρνούμαστε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε κιόλα ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τον ίδιο τον πολίτη και πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει ευκρινώς το σύστημα. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση για απορρίθμιση και απλούστευση του συστήματος, όχι μόνο για τι επιχειρήσει, αλλά πάνω απ' όλα για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κόχλιτσεκ από την ΚΟΕ και αντιπρόεδρος ταυτόχρονα της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω διάφορα απλά σχόλια. Καταρχάς, δεν είναι κακή ιδέα, πιστεύω, να ενοποιηθεί ο τύπος καταγραφής που θα χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους χάρτες μερικές φορές τα, καταφέρνουμε. Μπορούμε παραδείγματι να, τους, ε, να επεκτείνουμε το σύστημα όπως είναι για τις ε, άδειε κυκλοφορία των οχημάτων, για τις άδειε οδήγησης ή για το κτηματολόγιο, καταγραφή κτλ. Ωστόσο τα μητρώα αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα. Η ιδέα δεν είναι κακή όπως είπα, είναι καλή ιδέα. Κάποιος συνάδελφος είπε ότι δεν χρησιμοποιούν οι πολίτες, ιδιαίτερα οι πιο ηλικιωμένοι, την ε, ε, τεχνολογία της πληροφορίας. Εγώ προσωπικώς θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά ηλικιωμένο, αλλά χρησιμοποιώ τον υπολογιστή, όπως και ο πρόεδρος φαντάζομαι. Και στην ε, Τσεχική Δημοκρατία, ξέρετε, έχουμε αυτό που ονομάζεται... Όχι, εντάξει, νέο είστε μεν, αλλά είστε νέος εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε στην Τσεχική Δημοκρατία το λεγόμενο checkpoint, ένα σύστημα όπου έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα από την ίδια θηρίδα. Ε, είναι μια ιδέα που πιστεύω είναι χρήσιμη και μπορεί να επεκταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Τώρα αν αυτό μπορεί να γίνει και διασυνοριακά, μένει να εξεταστεί. Πάντα βέβαια είναι παρόν, ε, το, παρόν ο γλωσσικός φραγμός αλλά και η δυνατότητα αναγνωσιμότητας των εγγράφων, το ασύρματο δίκτυο ίντερνετ, το Wi-Fi είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο η κάλυψη δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι και δεν γνωρίζω για τις λοιπές χώρες. Εμείς στην Τσεχία είχαμε παραδείγματα τα τελευταία χρόνια καταγράψει σημαντικά κενά σε περιοχές όπου δεν υπήρχε σήμα του διαδικτύου. Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει να είναι ε, παρόν σε όλη την επικράτεια και αυτό βέβαια σαν σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτήν την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Θετικό ακούγεται. Πρέπει όμως και η ενιαία αγορά να γίνει πιο απτή, πιο πρακτική. Γιατί όταν ξυπνάει κάνει το πρωί δεν πάει να συζητήσει τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς, πάει στη δουλειά του. Επομένως έχουμε να κάνουμε με μια πρακτική λύση, με ένα πρακτικό βήμα αυτό θα εκπροσωπεί η ενιαία ηλεκτρονική θηρίδα. Και πρέπει τα δεδομένα που θα καλύπτονται να είναι επαρκή ταυτόχρονα. Καλό το Κοινοβούλιο σε νέες προσεγγίσεις με βάση τη γνωμοδότηση αυτή και σε σχέση με τον πολίτη ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί πολλές ε, υπηρεσίες ε, μέσω του Google ή του Facebook ε, το πράττει γιατί είναι πολύ αργό το σύστημα της διοίκησης. Το 2018 όπου θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα login για όλα τα κράτη-μέλη. Θα έχουμε την ανάγκη να εξασφαλίσουμε και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, άρα και τη σχετική νομοθεσία, ώστε να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία αυτά τα συστήματα. Βλέπουμε λοιπόν καλές ευκαιρίες για εξευρωπαϊσμό και των επιχειρησεών μας, αλλά και οι πολίτες χρειάζονται πιο καλή ψηφιοποίηση, πιο καλή ψηφιακή κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάλμος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την DigiConnect. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ επίσης για το καλωσόρισμα και το θετικό αντίκτυπο, τη θετική ανταπόκριση μάλλον σε αυτή την ανακοίνωση στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά ε, υπάρχει το θέμα της κινητικότητας ε, των ε, Ευρωπαίων πολιτών Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό απαιτεί τεράστιες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, αλλά δίνει και ευκαιρίες για να βελτιωθούν οι σχέσεις με τους συμπολίτε μας, όπως άλλωστε αναφέρατε. Θα διαπιστώσατε λοιπόν ότι αυτές οι αρχές που αναφερθήκαν και τις οποίες σχολιάσατε, ε, συνιστούν μια νέα εντελώς προσέγγιση σε ό,τι αφορά τι δημόσιε υπηρεσίε στο μέλλον, βασίζονται στον ανοιχτό χαρακτήρα, στη διαφάνεια, αλλά και στην διαθεσιμότητα των δεδομένων, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοικήσεων, διασυνοριακά, αλλά και απέναντι στου διάφορου εμπλεκόμενους φορεί, τους πολίτε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι δημόσιε διοικήσει θα μπορούν να χορηγήσουν ε, δημόσιε υπηρεσίε υψηλού επίπεδου. Είπατε ότι οι υπηρεσίε που σχετίζονται με τους πολίτε είναι λιγότερο παρούσε στην ανακοίνωση με τη διαθεσιμότητα των βασικών ψηφιακών στοιχείων που μας βοηθούν να προχωρήσουμε μπορούν να προχωρήσουν οι ποιοτικέ δημόσιες υπηρεσίες και για τους συμπολίτε μας. Ε, πολλά βεβαίως αφορούν τις επιχειρήσεις, αλλά κάποιες πρωτοβουλίες ε, που δημιουργούν, παραδείγματο χάρη, ε, ε, τις ενιαίες για την πληροφόρηση όπως το e-justice, τη δικτυακή πύλη e-justice, όλα αυτά μπορούν να διευκολύνουν ε, τη δουλειά και των επιχειρήσεων αλλά και των συμπολιτών μας. Έχοντας κατά νου όλα αυτά τα στοιχεία, πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού ε, προς αυτό το όραμα της ανακοίνωσης. Ε, θα πρέπει να έχουμε τη συνολική εικόνα για να, στην ανακοίνωση αυτή που θα οδηγήσει τη μετατροπή της δημόσιας διοίκησης που θα οδηγήσει διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα ε, μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων. Μπορούμε λοιπόν να επιταχύνουμε αυτή τη μετάβαση τη διακυβέρνηση προ την ψηφιακή εποχή και για τι επιχειρήσει και για του συμπολίτε μα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Μπορείτε τώρα να πατήσετε το κουμπί. Πολύ ωραία. Η εισηγήτρια έχει το λόγο, η Αγγέλικα. Ναι, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται έχουμε ένα κοινό στόχο, μια κοινή προσέγγιση σε όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για μια καλή αλλά και ισχυρή γνωμοδότηση. Ε, προ ενημέρωση να σα πω ότι το σχέδιο γνωμοδότηση έχει σταλεί προ ε, μετάφραση στι 8 Σεπτεμβρίου Οπότε έως το 10 Ιανουαρίου θα, μπορούν, θα μπορεί να εξεταστεί. 17 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Των τροπολογιών. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν στο ίδιο πνεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο χρονοδιάγραμμα. Το σχέδιο γνωμοδότησης ε, θα εξεταστεί 12 Ιανουαρίου του 2017 βεβαίως. Οι τροπολογίες ε, θα πρέπει να υποβληθούν ε, έως τις 17. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε 28 Φεβρουαρίου και όχι 29 ευτυχώς. Και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ η ψηφοφορία στις 25 Απριλίου. Θα είμαστε λοιπόν εμείς έτοιμοι δύο μήνες πριν και πιθανότατα το θέμα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Αυτά για το σημείο 5. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και την εισηγήτρια και τους κοιόδους και τους υπόλοιπους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως να περάσουμε τώρα στο σημείο 6. Ο Επίτροπος Έτιγκερ θα είναι εδώ μαζί μας σε δύο λεπτά στις τέσσερις ακριβώς. Ναι, παρακαλώ. Έχετε κάποιο σχόλιο. Α, στη συζήτηση θέλετε να μιλήσετε, μάλιστα. Προς στιγμή νόμιζα ότι είχατε κάτι άλλο να μας πείτε. Δύο λεπτά διάλειμμα. Um, uh, uh, Ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γκίντερ Έτιγκερ σε αυτή την ασυνήθιστη ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι. Ο κύριο Έτιγκερ, κατά πάσα πιθανότητα, βρίσκεται ενώπιον μα για τελευταία φορά από αυτή την ιδιότητα, διότι έχει έρθει να μας ενημερώσει για μια υπόθεση παλαιότερη, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 και, και μετά από αυτή την επίσκεψη, κατά πάσα πιθανότητα στις επόμενες ημέρες, θα αναλάβει το ρόλο του Αντιπροέδρου και αρμόδιου για τον προπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους. Συζήτησε λοιπόν στο πλαίσιο του διαρθρωμένου δομημένου διαλόγου μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής και κύριε Επίτροπε ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τη γενική ενημέρωση για την υλοποίηση πλευράς της Επιτροπής του Προγράμματος για το 2016 αλλά και παλαιότερων από πλευρά σα γιατί μετά κάποιος άλλος θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Στην ψηφιακή πολιτική πολλές εξελίξεις έχουν εμφυλοχωρήσει φέτος, το γνωρίζουμε, πιο πρόσφατα μάλιστα με τη δημοσίευση της αναθεώρησης του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας νέος κώδικας για τις τηλεπικοινωνίες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε για όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα μια άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω κύριε Επίτροπε στην Επιτροπή Ήτρε και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να ξεκινήσει η συζήτηση. με Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ξεκινώντας, κυρίε και κύριοι, ξεκινώντα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ε, μεγάλη προσθεμένη αξία από τα ερευνητικά μας προγράμματα όσον αφορά την ψηφιακή ε, τεχνολογία το έχουμε παρουσιάσει αυτό με, τα μεγάλα, με τις μεγάλες εκθέσεις για τη ρομποτική, αλλά πέραν της ε, ρομποτικής ή της κρατικής ή της μικρο ή νάνο τεχνολογίας, θέλουμε ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι κανένα κράτος μόνο του δεν μπορεί να είναι αρκετά ισχυρό, ώστε να έχει την πρόοδο στην έρευνα και την ανάπτυξη που θα επιτρέψει που είναι απαραίτητη για την πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κανένα κράτος δεν είναι μόνο του αρκετά ισχυρό. Σε μια εταιρική σχέση όμως, εταιρική σχέση μεταξύ βιομηχανίας και πολιτικής, μεταξύ ορίζοντα 20, 2020 και κρατών μελών, έχουμε τη δύναμη, έχουμε την απαραίτητη ισχύ και το μέγεθος έρευνα, ε, είτε πρόκειται για την ε, ρομποτική, ε, όπου μπορούμε να έχουμε την πρωτοπορία και επικίνδυνο να χάσουμε την πρωτοπορία στην αγορά όπως την ανωτεχνολογία, να ενισχύσουμε τις προσπάθειες με τα κοινά σημαντικά προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών. Δεν χρειάζεται να συμπράξουν όλα ανεξαρτώ στα κράτη-μέλη. Τέσσερα, πέντε, έξι κράτη τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με έναν τομέα και ήδη εμπλέκονται σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν μαζί με την βιομηχανία ένα ευρώ της του ευρωπαϊκού προπολογισμού μπορεί να μεταφραστεί σε 5, 6, 10 ευρώ στις επενδύσεις αυτές. Αυτή είναι η προσθέμενη αξία την οποία εγώ υποστηρίζω στις ευρωπαϊκές ερευνητικέ εταιρικέ σχέσεις. Το hyper, high performance computing που θέλουμε μέχρι το 2020 να έχουμε προωθήσει εγγράφεται ακριβώς σε αυτό. Για το 2018 κυρίες και κύριοι ήμασταν ε, σε θέση να ε, διαθέτουμε τους έξι από τους 20 μεγαλύτερους και πιο αποδοτικούς ε, υπολογιστές στον κόσμο. Και τώρα έχουμε έξι των Αμερικανών που είναι πιο ισχυροί από του δικού μα και τρει των Ασιατών που βρίσκονται λίγο πολύ στο επίπεδο με, το δικό, με του δικού μα. Άρα λοιπόν χρειάζονται οι επενδύσει, όχι όμω επί 28, όχι σε κάθε κράτο, ε, σε τρία, τέσσερα, πέντε, ε, μαζί με τη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία για να προχωρήσουμε. Πρέπει να έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μα για να προωθήσουμε και να συγχρηματοδοτήσουμε τι προσπάθειε αυτέ, γιατί ορισμένα κράτη έχουν ήδη μπει σε συμπράξεις, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και μπορούμε να, τους να τα υποστηρίξουμε μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αν δεν το πράξουμε αυτό και σε όλες τις δυνατότητες που θα μπορούσαμε να έχουμε σχέση με τα big data, με, τα μεγάλα, με τις μεγάλες μέρες δεδομένων, θα βρεθούμε στην οπισθοφυλακή. Το ίδιο σε σχέση με τις υποδομές. Είχαμε ιδιαίτερη ενασχόληση κατά τη διάρκεια του έτους με το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την πρόταση για τα 700 GHz. Εδώ έχουμε να κάνουμε με σχέδια επέκτασης των ε, ψηφιακών υποδομέων έως το 2020 όπου εξετάσαμε διεξοδικά τι ανάγκες για μεταφορά δεδομένων θα έχουμε στις επόμενες δεκαετίες. Προσθέτοντας λοιπόν όλες αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν από κοινωνικά δίκτυα, upload, download, τηλεϊατρική, η IoT, η βιομηχανία του 4.0, τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, τα συνδεδεμένα ε, φορτηγά, την αυτονομή οδήγηση, την αυτοματοποιημένη οδήγηση κτλ. Έχουμε την εικόνα του μέλλοντος. Εδώ λοιπόν έχουμε προσδιορίσει τρεις βασικούς στόχους. Θέλουμε την επέκταση του κεντρικού σημείου ε, παραγωγής αυτής της δυνατότητας, σχολεία, δημόσια κτίρια κτλ. και την συνδεσιμότητα. Δεύτερον, οι μεγάλες αρτηρίες των μεταφορών μας, δεν πρόκειται για τους δεν πρόκειται για τους αυτοκινητοδρόμους, θέλουμε να είναι σε θέση να ε, έχουν επαρκή δυνατότητα μεταφοράς φορτίου, ψηφιακού, όγκου ψηφιακού και επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε την προσθέμενη αξία σε ακίνητα, είτε είναι κατοικίες, είτε είναι εμπορικά ε, κτίρια, είτε πρόκειται για υποδομές σταθερές, πρέπει πια να μιλούμε για το αν θα είναι σε online ή σε offline mode, εάν θα είναι ταχείας σύνδεσης ή όχι. Τα gigabyte λοιπόν χαράζουν το μέλλον. Αυτό είναι το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες το οποίο σας έχουμε ε, καταθέσει από το Σεπτέμβριο του 2016. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα έρευνας για το 4G με 700 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό που διαθέσατε εσείς, που μπορεί να συμβάλλει με ένα ποσό το οποίο πενταπλασιάζεται χάρη στις επενδύσεις της βιομηχανίας, της Γερμανικής Τελεκόμ, της Alcatel, της Nokia, πενταπλασιάζεται παραλαμβάνω εάν μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την πρωτοπορία του 4G. Μιλούμε για την υλοποίηση της πέμπτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας για το 2020 και μετά. Και εδώ έχουμε τα 700 GHz, GHz ως ε, ευρύτητα φάσματος και έτσι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε έναν και δύο ακόμη τριμερείς διαλόγους μέχρι τα Χριστούγεννα ε, πιστεύουμε ότι η λύση μπορεί να βρεθεί σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ε, πρόταση αυτή. Έχουμε και τη στρογγυλή τράπεζα των ρυθμιστικών αρχών που αυτή τη στιγμή ε, απαρτίζουν ένα δίκτυο διαλόγου περισσότερο παρά αρρύθμισης, παρά νομοθεσίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε όμως την πολιτική φάσματος χάρη στον καλύτερο συντονισμό αυτών των ρυθμιστικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και σε σχέση με το φάσμα και την, ε, την ευρύτητα του φάσματος πιστεύουμε ότι χρειάζεται καλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός. Και εδώ η νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία. Ένα πλαίσιο ρυθμιστικό πιο σύγχρονο, πάνω απ' όλα ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να κινητοποιήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις. Ξεκινούμε με 500 δισεκατομμύρια ευρώ σαν πρόβλεψη για τις πρώτες φάσεις, είτε πρόκειται για την ή ε, να ή άλλο, είτε πρόκειται για το 5G και πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα 10 με, 15, με 20% της συγχρηματοδότησης, ιδιαίτερα για την, περίοδο, για την περιοχή της Υπέθρου ή τις γεωργικές περιοχές, εκεί όπου ίσως να μην είναι τόσο ελκυστική μια επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ με την εθνική, την περιφερειακή, την τοπική υποστήριξη και τα σχετικά ταμεία και βέβαια τα ευρωπαϊκά προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΤΣΕ ή το, τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συμπληρώσεις της χρηματοδότηση. Πριν από 1,5 χρόνο ξεκινήσαμε τον δομημένο διάλογο με τη βιομηχανία 4.0 μέσα από την ε, πλατφόρμα IoT. Έχουμε 10 ή 11 πλατφόρμες σε, όλη την Ευρώπη σε εθνικό επίπεδο. Στη Γαλλία, Φερρυπίν, στις κάτω χώρες με το Smart Vectoring, ε, το Catapult της Βρετανίας, το Industry 4.0 της Γερμανίας. Σε μια από κράτη λοιπόν όπου ενθαρρύναμε και ξεκινήσαμε με διασκέψεις την ίδρυση αντίστοιχων, ε, αντίστοιχης πλατφόρμας και ε, με συμμετοχή του κράτους αλλά και με συμμετοχή του κλάδου της βιομηχανίας. Και έτσι μπορέσαμε να ιδρύσουμε την πλατφόρμα που συνενώνει όλες τις πλατφόρμες για να συζητήσουμε ποια είναι τα θέματα που μπορούμε καλύτερα να εξυπηρετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε για παράδειγμα την κυβερνοασφάλεια. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα μόνο ενδεικτικά. Η κυβερνοασφάλεια λοιπόν, η ασφάλεια των δεδομένων, η ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών με την εκκίνηση ενός ε, ε, συνόλου προδιαγραφών για την ασφάλεια των ε, ψηφιακών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί θα αποδώσει καλύτερα. Και πρέπει να δούμε τις επενδύσεις σε υλικό και λογισμικό με πιστοποίηση από ανεξάρτητες ελεκτικές αρχές και μια σήμανση ευρωπαϊκή, επισήμανση μάλλον ευρωπαϊκή, μια ετικέτα ευρωπαϊκή. Επίσης το cloud, το νέφος λέει το ψηφιακό ή υπηρεσίες πληροφορικής μέσα από την κυβερνό ασφάλεια που μπορούν να αναπτυχθούν και να καταστούν παράγων της αγοράς, παράγων σημαίνων για την αγορά. Οι προδιαγραφές επίσης έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε 25 ε, διαφορετικές γλώσσες στην Φαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται όμως να έχουμε 28 διαφορετικούς μηχανισμούς μετάφρασης, μηχαν, ε, μηχανές μετάφρασης. Έχουμε πολλές εταιρείες, ε, την Volkswagen, την IBM, τόσες άλλες οι οποίες παράγουν υπηρεσία ε, στα 28 κράτη με διαφορετικά σημεία εγκατάστασης, αλλά δεν χρειάζεται τα μηχανήματα αυτά να μιλούν 25 ε, διαφορετικές γλώσσες ή ανάλογα με το κράτος στο οποίο βρίσκονται. Πρέπει να έχουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ τους και αυτό θα μας βοηθήσει να προσφέρουμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία για να μην έχουμε τον κατακαιρματισμό του, προσφερόμενου προϊόντος. Και τρίτον, οι περαιτέρω ψηφιακές υποδομές σε ένα δεύτερο διάλογο που θα, όπου θα προεδρεύσω εγώ, το Connecting Task, η οικονομία της τηλεπικοινωνίας πρέπει να συνεργαστεί. Αυτό θέλουμε να δείξουμε με τη βιομηχανία. Οι τηλεπικοινωνίες, οι επιχείρησεις των τηλεπικοινωνιών μέχρι τώρα έχουν οργανώσει την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων από το αυτό στόμα του ενός αυτή του άλλου, από το σημείο Α στο σημείο Β, με το σταθερό ή το κινητό δίκτυο. Ε, στο μέλλον όμως θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσουν και τη μεταφορά δεδομένων, το flow of data, σε όγκους όλο και μεγαλύτερους που σε πραγματικό χρόνο θα φτάνουν στον στόχο τους, ε, στο στόχο τους τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα χωρίς εκτεταμένη συνδεσιμότητα με υψηλή ποιότητα ε, και απόδοση σύνδεσης δεν μπορούν να υπάρξουν και η κινητή μας τηλεφωνία ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, γίνεται κατά τρόπον ώστε να ε, έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Κάποια κράτη έχουν μείνει πίσω, πρέπει ακόμα να προχωρήσουν το 3G στο 4G. Αν θέλουμε όμως να είμαστε στο 5G έτοιμοι όλοι ταυτόχρονα, τότε ένας αυτοκινητόδρομος φέρει ε, από το μόναχο στο Βουκουρέστι που θα παρακολουθεί τη ροή και του Δούναβη θα επιτρέπει ε, μια κάλυψη τέτοια που θα δίνει δυνατότητα και για αυτόνομη οδήγηση. Χωρίς αυτή όμως την κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων δεν μπορούμε να έχουμε την αυτόνομη οδήγηση και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κανένα κενό. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε ένα, μια ενιαία πολιτική φάσματος ευρωπαϊκή και στο διάλογο συνδέοντας τα αυτοκίνητα Connecting Cars έχουμε και τον παραγωγό της τεχνολογίας και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και την τεχνολογία, τη λυπή που πρέπει να συνομιλούν κατά τρόπο ώστε να μην μείνει κανένα απολύτως κανένα κενό. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε μια απόλυτη κάλυψη για κάθε δρόμο του 5G ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Ένα Ρενό του, 2017 ένα BMW του 2017, όταν το αγοράζει καλή, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι μπορεί να κυκλοφορήσει με απλό, απόλυτη αυτονομία, χωρίς κανένα λάθος στην κάλυψη του δρόμου. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν χωρίς κανένα κενό καλύπτονται τα οδικά μας δίκτυα από το 5G. Ζητήματα ε, η πετιότητα συμβα, συμβατικής ευθύνης και το έξω εξωσυμβατικής ευθύνης πρέπει να καλυφθούν επίσης ε, οι εξαιρέσεις που μπορεί να αφορούν κάποιους δρόμους όλα αυτά έχουν να κάνουν με την οργάνωση του 5G και θα ήθελα να αφαιρθώ στην ανακοίνωση που θέλουμε να δημοσιεύσουμε τον Ιανουάριο για την οικονομία ελεύθερης ροής δεδομένων για την ελεύθερη ροή των δεδομένων λοιπόν πέραν των συνόρων στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για θέματα που αφορούν τη φορολογία, την ασφάλεια, την αστυνομική νομοθεσία μεταξύ των κρατών, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να καταρρύψουμε τα υφιστάμενα αυτή τη στιγμή από το ένα κράτος στο άλλο εμπόδια. Ιδάλλως δεν μπορούμε να έχουμε ενιαία αγορά. Αυτό το free flow of data λοιπόν που μπορεί να συναντάει έως και 50 διαφορετικά εμπόδια, πρέπει να ε, εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα να προβλέψουμε και μελλοντικά ενδεχόμενα προσκόμματα που μπορεί να προκύψουν από τις εθνικές νομοθεσίες. Ε, στην ε, οικονομία των δεδομένων έχουμε πολύ συναρπαστικά ζητήματα αστικού δικαίου, το δικαίωμα πρόσβαση των δεδομένων, σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα, ποιος μπορεί να αξιοποιεί τα δεδομένα. Το αυτοκίνητο του μέλλοντος που θα έχει δεκάδες ε, αισθητήρε, είτε φωτεινότητας, είτε βροχής, θερμοκρασίας. Αυτά τα στοιχεία θα παίρνουν από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο, θα περνούν στο cloud, θα ε, την χάνουν κατεργασίας μαζί με τα αντίστοιχα δεδομένα χιλιάδων άλλων αυτοκινήτων. Θα ανήκουν στην Renault, στην Daimler, στην Bosch, στη Philips, στον κάτοχο του αυτοκινήτου, στον οδηγό ενδεχομένω του αυτοκινήτου πώς ρυθμίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Ή εάν ένας κινητήρας έχει ένα μικρό, μια μικρή ρογμή και στέλνει το μήνυμα ασθενό, αρρωσταίνω, διορθώστε με. Σε ποιον θα πάνε τα δεδομένα, θα πάνε στην Daimler, η Daimler θα το κρατάει, θα μπορεί να ε, κυκλοφορεί σε αυτή η πληροφορία, θα υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα και την αξιοποίησή του ή μόνο για ορισμένους θα είναι διαθέσιμα. Αυτά είναι τα ερωτήματα του μέλλοντος. Από την 1η Δεκεμβρίου θα ασχοληθούμε με ε, την διαμόρφωση της αγοράς της ψηφιακής για το μέλλον σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους εταίρους γιατί βλέπουμε ότι στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο χάνουμε 180 ειδικούς της πληροφορικής από το υψηλότερο επίπεδο. Καθένας από αυτούς που φεύγει χρειάζεται να αντικατασταθεί από έναν ή περισσότερους. Χρειάζεται κάθε χρόνο να έχουμε 180.000 νέους ειδικού. Δεν φτάνουν καν οι θέσεις που έχουμε στα πανεπιστήμια μας, στις, ε, στις ανώτερες σπουδές μπορούμε να προσφέρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουμε τον όγκο αυτό στην εκπαίδευση που θα καλύπτει και την ε, δυνατότητα για σπουδές της πληροφορίας, της τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής και βέβαια και η κατάρτιση και η πιστοποίηση και η μετεκπαίδευση των υφισταμένων εργαζομένων μας στους διάφορους τομείς ε, της τεχνολογίας. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια συμμαχία με τους ε, με τις ενώσεις των εργοδοτών, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τα κράτη-μέλη, ώστε να έχουμε κοινούς στόχους και η ψηφιοποίηση του κόσμου εργασίας να μην είναι εις βάρος των εργαζομένων μας, αλλά να τους βοηθά στην μετάβαση σε αυτή τη νέα μορφή εργασίας. Αυτά και μετά το 2017. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου κλείνοντα για, για την ιδιαίτερη ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι προτάσει μα. Σε άλλου τομεί τη πολιτική μπορεί να χάνονται και δύο και τρία χρόνια στι συζητήσει, αλλά στον ψηφιακό τομέα είτε πρόκειται για τα οπτικοακουστικά και τη σχετική ε, οδηγία για τι οπτικοακουστικέ υπηρεσίε. Δεν πρόκειται για τον εξυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών ε, ή είτε για οποιοδήποτε άλλο τομέα. Κάθε ε, στιγμή που χάνουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται ταχύτατα οι συνομιλίε και στο Κοινοβούλιο βέβαια και σε επίπεδο Συμβουλίου. Βλέπουμε ότι το κύρος μας και η ψηφιακή μας κυριαρχία, ευρωπαϊκή κυριαρχία, χάρη σε αυτό μπορούν να ενισχυθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων τώρα ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην ξεπεράσετε τα τρία λεπτά παρακαλώ για να μην βρεθούμε εκτός χρόνου. Από το ΕΛΚ τώρα η Αντιπρόεδρο Κοινοβουλίου κυρία Βαλέρν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πίτροπε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα λέει κυρία Βαλέαν. Σας ευχαριστώ για όλο το πακέτο το οποίο προσπαθείτε να προωθήσετε καθώς και για την προσέγγιση που σκοπεύετε να ακολουθήσετε, που είναι μια συνολική, σφαιρική προσέγγιση. Εδώ και καιρό ασχολούμαι με ζητήματα τηλεπικοινωνία σε αυτό το, σε αυτό το κοινοβούλιο και ποτέ δεν έχω δει μια προσέγγιση που να, έχει, ε, να, καλύπτει ένα τόσο ευρύ φάσμα και να έχει τόσο ευρύ αποδοχή από τους εμπλεκόμενου φορείς ε, και από τον κλάδο ουσιαστικά. Ο, ο ίδιος ο κλάδος λοιπόν θεωρεί ότι η πρότασή σας ανταποκρίνεται στα αιτήματά του και το πρώτο αίτημα, η πρώτη προσδοκία είναι η ασφάλεια και η σαφής κατεύθυνση. Είπατε, είπατε το 5G είναι το μέλλον, το είπατε με μεγάλη σαφήνεια και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό είναι το μέλλον, εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον κώδικα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, έχουμε έμφαση στην συγχρηματοδότηση ε, και αυτό είναι ενδιαφέρον και αυτό είναι καινούριο ε, έτσι ώστε να σπάσει αυτός ο κύκλος όπου χρειαζόμαστε επενδύσεις ε, και, να, πρέπει κάθε φορά να βρίσκουμε κίνητρα είναι μια σωστή προσέγγιση Θα θέλαμε να μας πείτε πώς οι ιδιωτικές επενδύσεις στη νέα αυτή γενιά την τεχνολογική θα επιβραβεύεται διότι είναι πολλές αυτές οι οι ε, επιχειρήσει που ενδιαφέρονται για τέτοιου επενδύσει. Τώρα, μια πολύ καλή ιδέα η οποία θα έχει ευρεία υποστήριξη είναι αυτό το πακέτο. Είναι βεβαίω τα, τα, κονδύλια, οι πόροι περιορισμένοι. Υπάρχει αυτή η ιδέα ε, του πολλαπλασιαστή, του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα αυτών των επενδύσεων και αυτών των ταμείων. Ε, θέλουμε να μας πείτε περισσότερα για αυτά. Επίσης, υπάρχει το θέμα της ελεύθερης ροής δεδομένων και της σχετικής ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί τον Ιανουάριο. Αυτά που είπατε, ότι θα πρέπει δηλαδή να απαλληφθούν τα εμπόδια για την ελεύθερη ροή των δεδομένων, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό ε, και εμείς θα υποστηρίξουμε αυτή την πρότασή σας έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα και ομαλά όπως είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Κομπούλα Νάτρη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ναι, καλωσορίζω αυτή την πρόταση ε, για το βασικό ε, διαδίκτυο, τη βασική πρόσβαση στο διαδίκτυο, η οποία να θεωρηθεί ε, βασικό δικαίωμα, η πρόσβαση, η προσβασιμότητα στις βασικές υπηρεσίες ίντερνετ είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Η, κοινωνία των gigabyte πρέπει να περιλαμβάνει όλους. Αναφερθήκατε στις δεξιότητες κύριε Επίτροπε, δεξιότητες ε, και για τη χρήση αλλά και για την δημιουργία καινοτόμων ε, τεχνικών. Το θέμα είναι πώς όλα αυτά θα επιτευχθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι νωρίτερα είχαμε θέσει κάποιους στόχους, τους οποίους τελικά δεν πετύχαμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη επιφυλακτικότητα από πολλά κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει απαραίτητη χρηματοδότηση ε, για να γίνουν αυτά που έπρεπε και μπορούσαν να γίνουν. Ούτε σε αυτόν τον παρόντα προπολογισμό τον ευρωπαϊκό υπάρχουν επαρκή σπόροι. Έχετε αναφερθεί από αυτού βεβαίω ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχουμε πει και εμεί ε, για τον Οριζόντα 2020 ότι είναι πολύ βασικό στόχος αυτός, αυτό που συμβαίνει σε πολλές χώρες και σε πολλές αγορές είναι ενθαρρυντικό. Εγώ παρακολουθώ το τι γίνεται στον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας, μόνο και μόνο ε, στην, ε, όσον αφορά τα κινητά δεδομένα, έχουμε αύξηση πάνω από 100% στην Πολωνία, 117% στη Λετωνία. Ε, ε, μικρές επενδύσεις, όχι πολύ μεγάλες, μικρές επενδύσεις που οδηγούν σε περισσότερα και φθηνότερα δεδομένα έτσι ώστε η κοινωνία των Gigabyte να γίνει πραγματικότητα. Βεβαίω χρειάζεται και η ενίσχυση των επενδύσεων, αλλά όταν υπάρχουν οι βασικέ δομέ, αυτό που πρέπει να, ενισχύσουμε την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες έτσι ώστε και οι καταναλωτές και η οικονομία να έχουν να αντιμετωπίσουν ελεύθερο ανταγωνισμό ε, και διαφάνεια. Πρέπει να έχουμε μια πιο φιλόδοξη ε, πολιτική σε αφορά το φάσμα. Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις ε, τη Κομισιόν ε, και του Κοινοβουλίου προ την κατεύθυνση αυτή, αλλά υπάρχει φυλακτικότητα από τα κράτη-μέλη. Το έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν. Θα ε, επανεξεταστεί και ο, ο σχετικό κανονισμό. Αυτό που έχει κάνει το Μπέρεκ σε επίπεδο συμβατότητα είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό στην άκρη σχέση με τι NRAs που λειτουργούν διαφορετικά. Οι λύσει για τι βάσει δεδομένων είναι σημαντικέ ε, για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, είναι όμω εξαιρετικά σημαντικέ και για την Ευρώπη και του πολίτε τη. Να πω ακόμα κάτι. Το θέμα τη κυβερνοασφάλεια. Στο έγγραφό μα είχαμε πει ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα τομέα ε, όπου πρέπει να επενδύσουμε. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που να ασχολείται με αυτό και να μην εμπιστευόμαστε πάντα τους, ξένου ξένους γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ECR. Ο κύριος Χένκελ, αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε Έτιγκερ, σας ευχαριστώ πολύ για την εντυπωσιακή σας παρουσίαση. Δείχνετε ότι και σε αυτή τη θέση επιτρόπου. Τα καταφέρατε τόσο καλά όσο και στην προηγούμενη και λυπούμε που κατευθύνεστε προς μια άλλη θέση. Αλλά με την ευκαιρία αυτή και στο τέλος αυτής σας της θητείας θα ήθελα να διατυπώσω μια ερώτηση για να μου δώσετε απαντήσεις. Ξέρετε ότι για χρόνια δραστηριοποιούμε στον τομέα αυτόν. Από το 80, το 90, το 2000, τα έχω ξανακούσει αυτά που μας είπατε. Διότι πάντοτε λέγαμε ότι πρέπει να προλάβουμε την υπεροχή των Αμερικανών, παλιότερα των Ιαπώνων. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν απορροφήσει χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου χωρίς αποτέλεσμα όσοι βρίσκονται εδώ ίσως να μην θυμούνται ακόμα τα ονόματα εκείνων των περίφημων προγραμμάτων, αλλά εγώ τα θυμάμαι, το ΕΣΠΡΙ, το ΕΒΡΙΚΑ, προγράμματα τα οποία είχαν ε, θεσπιστεί προκειμένου να προλάβουμε την πρωτοπορία των Αμερικανών ή των Ιαπώνων. Δεν τα καταφέραμε και μάλιστα υπήρχαν ε, τότε ακόμα οι Νίξτορφ, οι ICE, οι Ολιβέτη, οι Μπούλ, οι Φίλιπς, οι Τόμσον, οι Έριξον, οι Άντλερ, ε, εταιρείε ευρωπαϊκές υπολογιστών που όλες έχουν φύγει. Δεν έχουν ε, μείνει. Δεν έμεινε καμία εκτός από αυτές που μείνανε χωρίς την υποστήριξη του Ευρικά ή άλλων προγραμμάτων. Αν λοιπόν θέλουμε να κοιτάξουμε ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας οι κύριοι, η Microsoft, η Google, η Apple, το Facebook, το Twitter, δεν έχουν καμία σχέση με κρατικές επιχορηγήσεις. Και έχω να δείτε πόσο τα εξή βασικά ερωτήματα. Πρώτον, δεν θα ήταν σκόπιμα σκόπιμο πρώτο να κοιτάξουμε γιατί είχαν τέτοιο κόστος και τόσο μικρό ποσοστό επιτυχίας τα παλαιότερα αυτά προγράμματα. Γιατί απέτυχαν τόσο παταγωδός. Και δεύτερον, Πώς πιστεύετε, πού στηρίζετε την πίστη ότι μπορείτε με τα νέα αυτά προγράμματα εσείς ο διαδοχός σας επιτρόπος να έχετε καλύτερη επιτυχία. Uh, thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χένκελ. Η κυρία Μάισνερ από την Άλντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Έτσιγκερ, εκ μέρου των φιλελευθέρων. Τα όσα μα είπατε έχουν να κάνουν θέματα πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Τα γνωρίζουμε όλοι. Ήδη έχουμε μπει πια στην ψηφιακή εποχή. Και μπορώ να είμαι εγώ, αντίθετα από τον κύριο Χένκελ, πιο αισιόδοξη, γιατί πιστεύω ότι έχουμε σε πολλά κεφάλαια εισαγάγει την ψηφιοποίηση ριζικά έχει αλλάξει η ζωή μας, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερες ευκαιρίες, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε αν μπορούμε να τηρήσουμε τους ρυθμούς της ανάπτυξης. Και πρέπει να κοιτάξουμε εάν όλα αυτά που έχουμε κάνει μπορούν να φέρουν αποτελέσματα αρκετά γρήγορα από την προηγούμενη περίοδο με, το, με τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη τα 15 εκατομμύρια που είχαμε για την ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιακή οικονομία διαθέσει με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή οικονομία 9,2 ενώ τώρα νομίζω ότι είναι κάπου ε, πολύ λιγότερα τα ποσά ε, δεν ε, βλέπουμε να φέρουν αποτελέσματα θέσεις εργασίας και για την Ήπεθρο που έχει πολύ μεγάλη σημασία να δραστηριοποιηθούμε, για τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, για το sharing υπόνομη, όπου χρειάζονται πάντοτε οι υποδομές. Και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Από τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή βλέπετε αρκετή φιλοδοξία στην συγχρηματοδότηση των έργων. Βλέπετε να διατυπώνονται ε, προτάσεις για το ΕΤΣΕ ή για το Connecting Europe Facility ή βλέπετε να καθυστερούμε ακόμη. Βλέπετε κάποια σημεία στα οποία χρειάζεται να επιταχύνουμε το βήμα. Μπορείτε να μας αντοπίσετε κάποιους τομείς. Επίσης, λέτε ότι θα πρέπει να τυποποιηθούν οι γλώσσες των υπολογιστών, των μηχανών το ακολουθούν αυτό τα κράτη-μέλη. Φαντάζομαι ότι μάλλον η Αγγλική θα έχει επικρατήσει από διάφορε συζητήσει. Έχω αντιληφθεί πόσο δύσκολο είναι να συμφωνήσει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία και μόνο γλώσσα. Επίση για το connecting cars και το platooning ε, που αναφέρατε. Το γνωρίζω και από την Επιτροπή μου οι υποδομές για το Connecting Europe Facility έχουν σαν στόχο να, εισαγάγουν, να διευκολύνουν την και αυτή της νομοθεσίας με του συντονισμού του ΕΣ λοιπόν για τους αυτοκινητοδρόμους των μεταφορών ε, και τις υποδομές. Τι επαφές έχετε, μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί. Και μια πολύ στομή ερώτηση για τα δεδομένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Φαντάζομαι ότι έχετε στενή επαφή και συνεργασία με τον ε, υπεύθυνο για την προσέγγιση των προσωπικών δεδομένων, γιατί αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί. Και κάτι ακόμη από την επικαιρότητα των τελευταίων ημέρων, γιατί βλέπουμε σε εφημερίδε και ειδικότερα το Σπίγκελ να λέγεται ότι υπάρχουν προοπτικέ για νέε θέσει εργασία, αλλά χρειάζεται και αλλαγή ε, στην, στην ιεραρχία καλύτερα, στη διαχείριση των επιχειρήσεών μα και των ε, μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Ε, τι επαφές έχετε μαζί τους λοιπόν. Ευχαριστώ Γιάβορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε σήμερα. Καταρχάς, στις 18 Μαΐου φέτος ταξιδέψατε με ιδιωτικό τζέτ στην Ουγγαρία. Από ό,τι είπανε διάφοροι εκπρόσωποι λόμπι κτλ. Πάντως, δεν αναφέρθηκε στα προσωπικό σας ε, ε, blog. Όμως ε, δεν ενδιαφέρεστε για την ψηφιακή αγορά. Ο πρόεδρος Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που είναι υπό έρευνα. Δεν είναι θέμα της δικής μας συνεδρίασης σήμερα. Ξέρετε, η δημοκρατία είναι κανόνες και θεσμοί. Δεν είναι σήμερα αυτό το θέμα της, της συζήτησής μας. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν ε, η σχέση του κυρίου Μάγκορ με την ψηφιακή αγορά. Οπότε σαφώ σχετίζεται με την ψηφιακή αγορά πρώτον και κύριον και δεύτερον ποτέ παλιότερα δεν είχαμε την εμπειρία, δεν είχα την εμπειρία του περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης ενός ευρωβουλευτή από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής. Η ερώτησή μου πιστεύω ότι σχετίζεται με την, ε, το θέμα της ψηφιακής αγοράς και θα ήθελα να συνεχίσω αν μου επιτρέπετε. Μα δεν είναι εδώ ο χώρος να, να θέσετε τέτοιες ερωτήσεις και να απαντήσετε, γιατί έχουμε προετοιμαστεί για τελείως διαφορετική κατάσταση. Ξέρετε, ε, θα πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες τους δημοκρατικούς. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση ε, που ε, θα γίνεται στην Επιτροπή και ο Πρόεδρος Γιούνκερ είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα. Παρακαλώ λοιπόν αφήστε το κατά μέρος και θα αρχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα που έχουμε στην ημερήσια μας διάταξη. Γιατί είπαμε ότι το θέμα μας είναι αυτό που έχετε μπροστά σας και το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω ωστόσο να πω ότι αυτό που λέω σχετίζεται στενά με το πώς αντιμετωπίζει την ψηφιακή την ατζέντα για την ψηφιακή αγορά ο κύριος Έτιγκερ. Πώς έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που σχετίζονται ή όχι με την ψηφιακή αγορά. Πρόκειται για την ε, λογοδοσία του, για την εργασία του ως Επιτρόπου αρμόδιο για την ψηφιακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε λες και δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Σαφώς και δεν θέτω ερωτήματα σε σχέση με, αυτό το με θέματα που δεν ε, άπτονται του θέματος ψηφιακής αγοράς. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς είναι οι επαφές του με κάποιον που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και ε, ε, δεν σχετίζεται με την ψηφιακή αγορά, ενώ η Ουγγρική κυβέρνηση λέει πως έχει μια ε, σύμβαση για συμβουλευτικές υπηρεσίες με τον κύριο Μάνκορ και συμπεριλαμβανόμενε της οργάνωση της σύσκεψης στην οποία εσείς συμμετείχατε και που σχετιζόταν με το μέλλον του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο του μέλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω. Ποιο έχει δίκιο, η Ουγγρική κυβέρνηση που λέει ότι ο κύριο Μάγκολ ενδιαφέρεται για την ψηφιακή αγορά. Μα αγαπητέ συνάδελφε, διακόπτει ο πρόεδρο. Η δημοκρατία λειτουργεί επί τη βάση θεσμών και διαδικασιών. Μα είναι μια ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Δεν είναι μέσα στη διαδικασία μας, ε, στον κανονισμό μας, να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Παρακαλώ λοιπόν να μείνετε εντός θέματος. Ναι, ναι, και εσείς μπορείτε να πάρετε το λόγο, αν το θέλετε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέτω μια ερώτηση σε σχέση με μια επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου στις 18 Μαΐου στην, ε, στην Ουγγαρία. Και νομίζω πως είναι σημαντικό και για τη δική μας Επιτροπή να δούμε ξεκάθαρα πώς μετέβει σε αυτήν την σύσκεψη για την ψηφιακή αγορά και το μελλοντικό αυτοκίνητο και αν αυτό είναι σύμμορφο με τον κανονισμό που αφορά τους επιτρόπους εν γέννη. Μα δεν είναι εκτός ενδιαφέροντος ε, της ε, ψηφιακής ε, αγοράς. Κοιτάξτε, η Επιτροπή Συντα... Συνταγματικών Υποθέσεων είναι αρμόδια στο Κοινοβούλιο για τέτοια θέματα και μπορούμε να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα στη Συνταγματική Επιτροπή και ανοιχτά. Όπως θα θυμάστε στις ακροάσεις μας, πριν από δυόμιση χρόνια επίσης ανεφέρθη από κάποιους, νομίζω από κάποιον σοσιαλιστή, κάτι σχετικό με ερώτηση προς κάποιον άλλον και παρεπέμφθη στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Αυτό είναι όλο. Παρακαλώ λοιπόν συνάδελφε, μείνετε στο θέμα. Εάν δεν θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση σχετική με το θέμα μας, παρακαλώ ολοκληρώστε για να περάσουμε στον επόμενο μιλητή. Ναι, έχω διάφορες ερωτήσεις και θα ήθελα να σας ζητήσω να καταγράψετε ότι η Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για την ερώτησή μου που ρωτά αν ο Επίτροπος συναντά εκπροσώπους ε, ομίλων ή λομπίστες που ε, ασχολούνται με την ψηφιακή αγορά και ότι δεν μου επιτρέπεται να θέσω την ερώτηση απευθεία στον Επίτροπο, ο οποίος έχει έρθει σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση. Ναι, έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία και παρακαλώ να τηρήσετε τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό, συνάδελφε. Λοιπόν, λοιπόν πάμε στο στον επόμενο μιλητή ο κ. Κόχλιτσεκ από την ΚΟΕ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερώτημά μου δεν σχετίζεται με κάποια ιδιο... κάποια ταξίδια ή επιχειρηματικά ταξίδια του Επιτρόπου. Σας ευχαριστώ, κύριε ε, Επίτροπε, για την ε, εισαγωγική σας, εισαγωγική παρέμβαση. Διαπιστώνω ότι εσείς βεβαίως ασχολείστε με την ψηφιοποίηση. Ποια κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτό το κοινό project. Είπατε 5 με 8 χώρες. Δεύτερον, ε, οι νανοτεχνολογίε. και αυτέ αποτελούν μέρο ε, των ζητημάτων ε, που αναφέρατε. Είναι το μέλλον η νανοτεχνολογία. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε στον τομέα των νανοτεχνολογιών. Τρίτον, η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να αποτελέσει θεμελιώδης δικαίωμα των πολιτών της Ευρώπης. Και θα πρέπει να έχουμε πλήρη κάλυψη, όχι μόνο των αστικών περιοχών. Είναι ένα θέμα το οποίο διαπιστώνουμε ότι είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή. Η κάλυψη δεν είναι 100% αυτή τη στιγμή, δεν είναι στο 100% και θα πρέπει ε, σε επίπεδο κρατών μελών να βελτιωθεί η κάλυψη για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Βλέπετε να υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης. Τώρα, οι διασυνοριακές υποδομές οι RTMS, οι σειροδρομικές υποδομές. Να ένα καλό παράδειγμα ε, διασυνοριακό. Ή το e-call, επίσης ένα πολύ καλό σχέδιο υποδομών. Ή ε, η οδική πλοήγηση, ε, παρότι υπάρχουν βεβαίως ακόμα ελλείψεις και κενά. Ένα άλλο ζήτημα Όταν πάτε σε ένα γκαράζ με το αυτοκίνητό σας, δεν αντικαθιστάτε μόνο ένα εξάρτημα, αντικαθίσταται ε, ένα πολύ πιο μεγάλο κομμάτι του αυτοκινήτου και αυτό ε, δημιουργεί πολλά ε, απόβλητα, αν θέλετε. Και αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε. Πιστεύετε ότι ο νέος κώδικας ε, θα είναι στα αγγλικά ή σκεπτικοπεύετε να ακολουθήσετε μια άλλη οδό. Μάλιστα, τέλος ερωτήσεων εκ των πολιτικών ομάδων. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε κύριε Επίτροπε εν συντομία, διότι έχουμε ακόμα 12 ομιλητές και πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει σε ένα τέταρτο. Οπότε θα ζητήσουμε ένα λεπτό παρεμβάσεις στη συνέχεια να το γνωρίζετε για τις λοιπές παρεμβάσεις δηλαδή. Τρία λεπτά είχαν οι εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων. Πολύ σύντομα, αν μπορείτε, κύριε Επίτροπε, για να απαντήσετε στα ερωτήματα και στη συνέχεια θα πάμε στα υπόλοιπα. Για την κυρία Βαλαιάνη, οι απαραίτητες επενδύσεις για την οπτική, για την ή αλλού και το, το ευρύ φάσμα θα χρειαστούν για να πραγματοποιηθούν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ανοίξουμε το, τη δυνατότητα για το πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών στην ιδιωτική βιομηχανία κατά 80-90%. Επίσης οι συνεπενδύσεις, αυτό που λέμε co-investment, πρέπει να προχωρήσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Καλό είναι να γίνεται η κατάσταση υποδομής μία φορά, όχι με τέσσερα διαφορετικά σχέδια. Επίσης, ε, σκοπεύουμε να ζητήσουμε στο δυνατόν ταχύτερη έγκριση των ε, έργων, ε, γιατί έχουμε ένα τριψήφιο ποσό Ε, που περιμένουμε να εγκριθεί για την υποστήριξη μέση χρηματοδότηση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αν υπάρχει λοιπόν ζήτηση πρέπει να είμαστε θέση να αντιδρούμε ταχύτατα και να εξασφαλίζουμε τα σχετικά ποσά. Ιδιαίτερα για την Ήπεθρο μπορούμε να πούμε ότι το μέσον θα είναι εξαιρετική ευκαιρία για τον πολίτη, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται, να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον ένα δημόσιο κτίριο, είτε είναι το Δημαρχείο, είτε είναι το σχολείο, που θα του προσφέρει ταχύτατη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, αναφέρθηκε το Connecting Europe Facility. Βεβαίως, τα ενεργειακά δίκτυα, η αγωγή αερίου, οι ψηφιακές υποδομές ε, είχαν ε, ήδη προσφέρει προταθεί ως ιδέα και βέβαια οι οδικές ε, υποδομές και οι σιδηροδρομικές από το 2012 με τη δεύτερη επιτροπή Μπαρόσο. Είχαν περικοπεί τα ποσά από το Συμβούλιο στα 6 δισεκατομμύρια στο ψηφιακό τομέα όμως. Η συνάδελφος Νέλη Κρούς ε, είχε κάνει περικοπή στο 1 δις. Και το πρόβλημα με το έτσι είναι ότι αν έχουμε ένα χωριό με 3.000 μια μικρή πόλη με 3.000 κατοίκους. και ένα άλλο μέρος με πολύ πιο περιορισμένο αριθμό κατοίκων δεν ε, μπορεί να είναι αποδοτική η, η, η εγκατάσταση ίνας ή άλλου γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο και είναι πολύ μικρός ο αριθμός των συμβασλωμένων εκείνων δηλαδή που θα συνάψουν μια σύμβαση και άρα χρειάζεται κάποιο τύπου υποστήριξη χρηματοδότηση με προγράμματα ενισχύσεων είτε εθνικά, είτε περιφερειακά, είτε τοπικά. Εδώ λοιπόν το έτσι μπορεί να αποτελέσει ένα όχι τόσο πρόσφαρο, πρόσφορο ε, εργαλείο γιατί καλύπτει πιο πολύ την τεράστια ε, κλίμακα υποδομής και δεν μπορεί να αντισταθμίσει πολύ γρήγορα τις πρώτες απώλειες από την λειτουργία. Εμείς Προσπαθούμε μας με τα κράτη-μέλη να αναπτύξουμε συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για την αξιοποίηση των μέσων για την ψηφιακή υποδομή. Για το συντονισμό φάσματος πέραν των συνόρων αυτή περιλαμβάνεται στην πρόταση για τις τηλεπικοινωνίες. Δεν θέλουμε να θέσουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την πολιτική για το φάσμα. Ταυτόχρονα τα έσοδα από τις διάφορες επιλογές συχνοτήτων δεν θέλουμε να μπαίνουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αν και θα είχαμε και γι' αυτό κάποια επιχειρήματα. Αλλά ζητούμε το συντονισμό, ώστε το 5G εγκαίρως να διαδραματίσει το ρόλο του γιατί το 2G, το 3G, το 4G η Ευρώπη ήταν πάντα μπροστά στην ε, έρευνα και την ανάπτυξη. Στο rollout όμως της τεχνολογίας δεν έχουμε την πρωτοπορία. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε με το 5G μετά την Νότια Κορέα αλλά τουλάχιστον να συμπορευθούμε με άλλες περιοχές του κόσμου με το 2020 να είμαστε έτοιμοι για το rollout του 5G ώστε να μην καθυστερήσουμε, να μην υπολοιπόμαστε σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Για την κυβερνοασφάλεια, αυτές οι ΣΔΙΤ για την κυβερνοασφάλεια, μπορούν να ενισχύσουν την ε, ε, βιομηχανία της Ευρώπης για την κυβερνία, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Έχω ήδη εντυπωσιαστεί από διάφορες επαφές που είχα από παραγωγούς τέτοιου ε, τέτοιου δυναμικού κυβερνοασφάλειας. Η Ευρώπη είναι μπροστά, το έχουμε πει και νομίζω ότι με τις δίτα αυτές μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Και εδώ έχουμε ένα θεμελιώδη ζήτημα. Έρευνα θεμελιώδης ή έρευνα εφαρμοσμένη για την Ευρώπη. Εγώ ιδιαίτερα θέλω να μπορεί η βιομηχανία να μας δώσει τις συμβουλές, τις σωστές συμβουλές. 700 εκατομμύρια ε, από τον δικό σας προπολογισμό του 5G. Το πενταπλάσιο όμως θα το διαθέσει η βιομηχανία, ο κλάδος. Αυτό θα είναι και το κριτήριο για το κατά πόσον είναι αυτές οι ΣΔΙΤ ε, αποτελεσματικές και παραγωγικές. Το ίδιο για τη ρομποτική. Η ABB, η η Κούκα, η Siemens, όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν μπει στην προσπάθεια αυτή και λέμε ότι μπορούμε να παραμείνουμε πρωτοπόροι στη ρομποτική, όπως και πριν. Για την κβαντική έρευνα, τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα, η Γκρενόμπλη, η Λιόν, το Δέλφτ, το Ούλμ, το Μόναχο, είναι μέσα στα έργα, συμμετέχουν όλα τα κράτη και έχουμε σημαντική πολλαπλασιαστική δράση για το ευρωπαϊκό συμφέρον, για, τα, για τη μικρο και νάνο τεχνολογία και ηλεκτρονική. Ε, πέντε κράτη-μέλη συμμετέχουν. Η Αυστρία και το Βέλιο αυτή τη στιγμή κάνουν τις επαληθεύσεις και πάντοτε με γνώμονα είναι δυνατόν να λειτουργήσει ο σχετικός κλάδος για την παραγωγή. Γιατί αν δεν υπάρχει για την ανοτεχνολογία παραγωγικός ε, κλάδος, παραγωγική βιομηχανία, δεν θέλουμε να διαθέσουμε σε κάποιον άλλον την έρευνά μας, το αποτέλεσμα της έρευνάς μας. Άρα θέλουμε και ο ιδιωτικός κλάδος να προσφέρει ποσό ισόβαθμο, ε, ε, ισότιμο με αυτό το οποίο εμείς δίνουμε για την έρευνα ως επιδότηση, αλλά ταυτόχρονα και η ανάπτυξη να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος προστασία δεδομένων. Ε, στη φάση αυτή κάνουμε την, ε, τον εξυγχρονισμό της οδηγίας για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Ξέρετε ότι ε, στην κινητή ιδιαίτερα τηλεφωνία και γενικότερα μέτρο των τηλεπικοινωνιών γίνεται η προσαρμογή, είναι απαραίτητη μάλλον η προσαρμογή της σχετικής οδηγίας. Στις 11 Ιανουαρίου θα καταθέσουμε τις προτάσεις για, την, για τον εξυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας για το αν θα υπάρχει μία γλώσσα επικοινωνία των μηχανών για να αυτή θα είναι η αγγλική. Κοιτάξτε, καταρχά υπάρχει ανάγκη για την τυποποίηση με το Σέντο, τη ΣΕΝΕΛΕΚ, το ΕΝΤΣΙ και πολλά άλλα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με του πρωτοπόρου στη βιομηχανία, παρατηρούμε, εμεί, παρακολουθούμε και συντονίζουμε αυτέ τι προσπάθειε και αν δεν μπορεί ο κλάδο να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, τότε θα μιλήσουμε εμεί για επιβολή προτύπων ευρωπαϊκών από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πάντως, στα, στην επικοινωνία από το, με, το ενός μηχανήματος με το άλλο σε επίπεδο εργοστασίου πρέπει να είναι κοινή η γλώσσα. Γιατί πολλές φορές ήδη μέσα στον ίδιο όμιλο ε, ε, Παραγωγικέ εγκαταστάσει δεν βρίσκονται πια στην ίδια χώρα. Πρέπει όμω να επικοινωνούν μεταξύ του τα μηχανήματα ή σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγή πρέπει να μιλούν τα μηχανήματα. Έτσι λοιπόν ο αυτοματισμός τη γλώσσα που θα μιλούν τα μηχανήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτω του ποια θα είναι τα πρότυπα που θα επιλεγούν πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα και βέβαια αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια πρότυπα για το μέλλον που θα έχουν ρίζα ευρωπαϊκή. Οι πλατφόρμε και η ψηφιοποίηση μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη βάση για όλα αυτά. το Μάιο αλλά και πιο πρόσφατα το Νοέμβριο η παραμονή μου στη Βουδαπέστη είχε αποκλειστικά και μόνο τον στόχο της παρακολούθησης μιας ψηφιακής ή μάλλον της παρουσίας μου σε μια ψηφιακή διάσκεψη με ομιλία την οποία εκφώνησε εκεί η ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία που, που επενδύει στην Ουγγαρία, που παράγει ε, είτε Audi είτε είναι στο ψηφιακό κέντρο της Bosch ε, που προέρχεται από τη Στουτχάρτη όπως και εγώ, έχει παραγωγική μονάδα της Bosch στη Βουδαπέστη. Για λίγη ώρα πήγα εκεί γιατί ήθελα ακριβώς τα κράτη Βίζεγκρατ να, έχουν μια να αναγνωρίσουν μια προστιθέμενη αξία στον ψηφιακό κόσμο και να μην παραμένουν ευρωσκεπτικιστικά. Τα κράτη αυτά, άρα και η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακία και η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν σημαντικό ρόλο σε προστιθέμενη αξία με την αυτοματοποιημένη βιομηχανία και τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα να προσφέρουν ένα εξαιρετικό μέσον και μια εξαιρετική ευκαιρία για την συνεργασία στα μεγάλα αυτά σχέδια και επίσης είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας ενός διασυνοριακού τεστ για αυτόνομα η οδήγηση ή κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μόνο σε ένα κράτος. Θέλουμε από τη Νότια Γερμανία, μέσω της Αυστρίας, της Σλοβακίας, την Ουγγαρία, τη Σερβία, μέχρι και τη Ρουμανία να μπορούμε να κάνουμε μια διαδρομή που θα καλύπτει 5-6 κράτη-μέλη και με υποψήφιο κράτος βέβαια τη Σερβία, 6-7 διαφορετικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πέραν βεβαίως των ισχυών των κανόνων της οδικής κυκλοφορίας, πέραν αυτών, αυτών εξαιρουμένων δηλαδή, να έχουμε κανόνες κοινού που θα εξυπηρετούν την αυτόνομη οδήγηση. Γιατί αυτό μόνο μέσα σε ολόκληρη την Ήπειρο διασυνοριακά δηλαδή μπορεί να εξασφαλιστεί και όχι μέσα στα εθνικά σύνορα ενός κράτους. Η Ουγγαρία ήταν ο οικοδεσπότης ε, τον Μάιο και τον Νοέμβριο πάλι όπου έδειξαν αντίστοιχα προϊόντα, είχαμε τους εταίρους παρόντες. Υπηρεσιακή ήταν η επίσκεψή μου στην ε, Ουγγαρία για την πυρηνική ενέργεια, ενώ και εδώ και δύο χρόνια δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, μονόλεπτες ε, παρεμβάσεις τώρα. Αν μπορείτε και λιγότερο, 50 δευτερόλεπτα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι πρέπει να αξιολογούμε έναν επίτροπο για την δουλειά που κάνει στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου του. Πρέπει όμως να αναγνωρίσω ότι κάποιες δηλώσεις και κάποιες ε, κάποια ταξίδια πραγματικά αμφισβητούν το κατά πόσο είναι το ιδανικό άτομο για αυτή τη θέση. Λοιπόν, για την ενιαία ψηφιακή αγορά και τις τηλεπικοινωνίες, ε, για το πρώτο ήθελα να πω, ποια είναι η απόψή σα για το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ένα δικαίωμα ανταμοιβή για τους ε, παραγωγούς ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγουμε τις ζώνες αποκλεισμού αλλά δεν πρέπει να υπάρχει πολύ ακαμψία στην αγορά. Να βάζουμε δηλαδή κυρώσει σε κάποια επιχείρηση που δεν είχε προβλέψει ε, τις επενδύσεις προς το ρυθμιστή. Μάλιστα, πολύ καλά. Ευχαριστώ ο κύριος Μαλτά. 15 δευτερόλεπτα γίνεται. Ναι, θα προσπαθήσουμε ακόμα πιο σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μιλήσω για, την επίσκεψη στην Βουδαπέστη με το ιδιωτικό τσέτα αφού υπάρχει έρευνα εν εξελίξη. Κύριε Επίτροπε, σε οποιαδήποτε δημοκρατία όμω, θα σα είχαν υποχρεώσει ε, να παραιτηθείτε μετά τα ρατσιστικά και υβριστικά σα σχόλια. Αν ήσασταν Γερμανό υπουργό, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να μείνετε στη θέση σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν νομίζω να είναι αυτό το θέμα του δομημένου διαλόγου. Είπα στην αρχή τη συζήτηση. ότι συνεχίζεται ο διαστροτημένος διάλογος ε, για αυτό το πακέτο. Δική σας ευθύνη βέβαια να πείτε ό,τι θέλετε. Ο κ. Ραϊμόν έχει το λόγο. Ε, ναι, ευχαριστώ και από μένα μια σύντομη ερώτηση, κύριε Επίτροπε, διότι δεν είναι σαφέ πως μια εξέλιξη σε σχέση με την ανάληψη των καθηκόντων επιτρόπου για τον προϋπολογισμό ε, μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις περισσότερες. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Είναι ιστορικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό αναφέρει. Ε, υπάρχει σχετικό παράτημα το οποίο μπορούμε να σας εξηγήσουμε. Τώρα ο κύριος Μαραγκάλ έχει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, δεν είναι μόνο ευθύνη μας να θέτουμε ερωτήσεις, είναι και δικαίωμά μας, έτσι. Και έχω την εντύπωση ότι ο Επίτροπος Έτιγκερ είναι εδώ ως υπεύθυνος για την ψηφιακή ε, ατζέντα και Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να θέσουμε μια σειρά από ερωτήσει, να εκφράσουμε την άποψή μα ή την ανησυχία μα για οποιαδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή σχετίζεται με τι αποφάσει και τι πράξει του Επιτρόπου για την ψηφιακή ατζέντα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να δώσει εξηγήσει, κάτι που δεν έχει κάνει ω τώρα, ποιο ήταν το νόημα αυτή τη επίσκεψη στην Ουγγαρία, ε, την ε, επίσκεψη σε έναν ε, ηγέτη, σε έναν ε, επικεφαλής κράτους μέλους που να μείνει στην ατζέντα του, έτσι. Ποιο είναι το νόημα και πώς σχετίζεται αυτό με τα καθήκοντά του ως υπεύθυνο για την ψηφιακή ατζέντα. Και ακόμα αναμένουμε απαντήσεις. Αυτά. Ευχαριστώ ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή δουλειά σας ως Επίτροπος ε, για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ε, βεβαίως οι υποδομές σήμερα είναι αυτές ε, που δίνουν δυνατότητα στην κοινωνία μας, στην οικονομία μας να προχωρήσει στο μέλλον. Ένα ερώτημα και ακόμα δύο μικρά ερωτήματα. Πρώτον, πώς θέλετε να συνεργαστείτε με τους ε, ηγέτες ε, τους ε, εκπροσώπους μάλλον των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ε, εάν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο με την συμπέριληψη των 5G είναι σημαντικό για να μην υπάρξουν αποκλεισμένοι να υπάρξει ενεργή συμμετοχή της υπαίθρου. Πώς θα δημιουργήσετε κίνητρα για τις επιχειρήσεις, διότι από τις επιχειρήσεις εξαρτάται, όχι μόνο από, τους, από τα κονδύλια. Πρέπει να υπάρξουν σημαντικέ επενδύσει στον τομέα του 5G και κάτι τελευταίο για τα, κράτη-μέλη. Πρέπει να πάρθουν κάποιε αποφάσει ταυτόχρονα. Πώ θα συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη για να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρίφιν έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και για τα σχόλιά σα προηγουμένω για την πρόσβαση στην, στον ψηφιακό κόσμο που πρέπει να είναι βασικό ε, θεμελιώδε δικαίωμα. Ανησυχώ ότι αυτό δεν θα το πετύχουμε και ανησυχώ ιδιαίτερα για τα άτομα ε, που ε, βρίσκονται ε, έτσι οι δράση τους είναι μεταξύ δύο τομέων σε εθνικό, σε διακυβερνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, έχουμε και το, το χειμερινό πακέτο για την ενέργεια. Το θέμα της αποδοτικής κρίσης της ενέργειας είναι κρίσιμο. για οποιαδήποτε αύξηση 1% στις τη της ενέργειας ε, μπορούμε να βγάλουμε πολλού ανθρώπου από τη φτώχεια. Χρειάζεται έξυπνη διαχείριση τη ενέργεια, χρειάζονται κτίρια τα οποία να είναι φιλικά προ την αποδοτική χρήση ενέργεια. Πώ λοιπόν σκοπεύετε να πετύχετε την ε, απαλλαγή από τον άνθρακο και την στόχου γενικότερα τη Ενεργειακή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τοσενόφσκι έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ενέργεια που έχει αφιερώσει στην ψηφιακή ατζέντα. Συμφωνώ με τα όσα είπε σε σχέση με περισσότερες επενδύσεις για την έρευνα για την κυβερνοασφάλεια. Η δημόσια χρηματοδότηση είναι απαραίτητη σε αυτό το τομέα. Έχω μια ερώτηση ωστόσο. Μιλήσατε για την τυποποίηση της γλώσσας ε, στην ε, ε, ψηφιακή τεχνολογία. Εγώ ασχολούμαι με αυτήν ολόκληρη μου τη ζωή και είναι πραγματικά στο χώρο της ουτοπίας μια κοινή γλώσσα. Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να οριστεί από το interface. Αυτά τα ανομοιογενή συστήματα επικοινωνούν και αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ κρίσιμο γιατί ενώπιον μας έχουμε ε, το θέματα wifi, μικρά συστήματα. Ωστόσο αυτό θα είναι το πιο σημαντικό γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη διοίκηση, για τη διακυβέρνηση αλλά και για την, ένα ελεύθερο περιβάλλον. με υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού και ανεξαρτησίας. Η ερώτησή μου είναι, έχετε καμιά, ε, κάποια ιδέα για το πώς θα λειτουργήσει αυτό σε διοικητικό επίπεδο. Ε, Ο κύριος Μπουτικόφερ. Παρακαλώ ένα λεπτάκι. Μα ασφαλώς, Πρόεδρε. Αν και πρέπει να πω πως εκπλήσωμε για το ότι αφενός έχουμε ως Επιτροπή το καθήκον να τυπώσουμε έκθεση για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και από την άλλη μας δίνεται το πολύ ένα λεπτό για να μιλήσουμε. Νομίζω ότι είναι δυσανάλογος ο περιορισμός, παρότι είχα ζητήσει μάλιστα πολύ νωρί το λόγο. Στο χρόνο που μου μένει θα προσπαθήσω να διατυπώσω δύο σύντομε ερωτήσεις, κύριε Έτσιγκερ. Πρώτον, η βιομηχανία της Γερμανίας αποτελεί, ε, έχει μια αρχιτεκτονική αναφορά για τον τομέα του manufacturing, για την ψηφιοποίηση και συνεργάζεται στη βάση αυτή με το IIC για μια περαιτέρω εξέλιξη. Ωστόσο δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ενοποιημένη προσπάθεια για τον ίδιο στόχο. Πώς σκοπεύετε να το αλλάξετε αυτό. Δεύτερον, για τις ε, υποθέσεις Άικστρον και Κούκα, εσείς ο ίδιος συζητήσατε δημόσια τα θέματα αυτά, πώς δηλαδή ε, πραγματικά στολίδια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπορούμε να αποφύγουμε να πουληθούν σε ξένους. Πολύ σύντομα λοιπόν, πρακτικά, πέραν κάποιων ε, κρίσιμων, ή επικριτικών παρατηρήσεων που μπορεί να διατυπώσατε. Δεν έχω τελειώσει την πρότασή μου, Πρόεδρε. Τι μπορείτε να κάνετε, υπάρχουν προσπάθειες, ώστε, γιατί είχατε αναφέρει Προνόητερα αφήσατε 1 και 45 το συνάδελφο. Αφήστε μου και εμένα 1 και 20 δεύτερα. Τι κάνετε λοιπόν προκειμένου το σύστημα το αμερικανικό, ο πρόεδρος διάκοψε, διάκοψε τον Μητρέ. Κοιτάξτε, ο συνάδελφος ο κύριος Γιάβορ έχασε τρία λεπτά χωρίς να διατυπώσει καμία σοβαρή ερώτηση για, το θέμα, για θέματα του δομημένου διαλόγου. Να είστε δίκαιος απέναντι σε μένα κύριε πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπιτικόφερ ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω στον τομέα του ε, wholesale roaming, του hidden roaming που έχουμε επίσης να συζητήσουμε γιατί έχετε ε, υποσχεθεί roam like at home να έχουμε δηλαδή περιαγωγή όπως ακριβώς και στον, ε, στο χώρο κατοικίας όπως και στην οικία χώρα. Ε, μπορεί να παραμείνει αυτό μέσα σε εθνικά σύνορα η τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, αν μείνουν σε εθνικά σύνορα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ψηφιακή εσωτερική αγορά, γιατί δεν μπαίνουν μέσα σε αυτή την ε, εσωτερική αγορά οι επιχειρήσεις των ε, τηλεπικοινωνιών και βέβαια αυτό δεν επιτρέπει και στις αντίστοιχες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Με 5G, με ψηφιακή ε, αγορά, με τα με συνθήκες ισοδύναμης πρόσβασης, ισότιμης πρόσβασης για τα 28 κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά, αντίστοιχα με τις ψηφιακές υπηρεσίε που έχουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαφοζέρ. Πολύ σύντομα, ευχαριστώ. Εγώ δεν σα ε, κατηγορήσω για τα ταξίδια στην Ουγγαρία. Νομίζω πω ε, κάτι τέτοιο δεν έχει εδώ χώρα. Αυτό που ζητώ από έναν επίτροπο είναι να είναι καλό επίτροπο καταρχά. Εγώ έχω ερωτήσει να σα θέσω. Γιατί στο ευρωπαϊκό cloud δεν ρωτήσατε την πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία, την OVH, για την ηλεκτρονική τεχνολογία, γιατί δεν προσπαθήσατε να έχετε απόλυτη ε, κυριαρχία στο λογισμικό και στο hardware, ειδικά για τους μικροεπεξεργαστές που έχουμε με το STM ακόμα. Γιατί δεν ακούσατε για το ευρωπαϊκό cloud τους ε, βιομήχανους που είναι 100% Ευρωπαίοι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζοχίνιο. Κύριε Επίτροπε, εγώ Συνυπογράφω την απορία, τις απορίες σε σχέση με το ειδική δική σας συμπεριφορά εκτός της ψηφιακής ατζέντα, αλλά έχω και δύο ερωτήσεις για την ατζέντα σας. Τα μοντέλα πρόσβασης ε, τα συζητήσατε, μιλήσατε για το στίχημα για τα 5G, για την πρόσβαση, καθολική πρόσβαση για όλους, ανταγωνιστική στο ίντερνετ και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Όμως η πρόσβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει ε, μόνο για ένα συγκεκριμένο σύστημα γιατί αλλιώς είναι αμέσω ε, ξεπερασμένα, πεπαλαιωμένα. Πώς λοιπόν θα δημιουργήσουμε τα θεμέλια για την ψηφιακή ε, διακυβέρνηση της Ευρώπης ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στη νέα φάση του ψηφιακού κόσμου. Δεύτερον, τι πιστεύετε για τις ταυτότητες που ορίζονται με βάση τη ζήτηση, δηλαδή από την, ε, με βάση την ικανοποίηση των πολιτών, ε, όχι με βάση την προσφορά, με βάση τη ζήτηση που κάνει και η βορειοαμερικανική αγορά. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής στον καταλογό μου είναι η κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τη δράση σας, την πολύ θετική σας δράση για τη δημιουργία αυτή της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Πριν να φτάσετε μόλις, συζητήσαμε το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η αρχή που αναφέρεται ε, εκεί είναι πολύ θετική, μάλλον οι αρχές που αναφέρονται είναι πολύ θετικές και ιδιαίτερα για τους πολίτες, αλλά και για τις εταιρείε μας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες. Για να λειτουργήσει αυτό, αν γέννη επίτροπε, ε, δηλαδή η ψηφιακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και για να υπάρχει εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ποια εργαλεία ε, για την ενίσχυση της ασφάλειας. Μιλήσατε για ετικέτες και πιστοποιήσεις. Μπορείτε να μας ε, αναπτύξετε κάπως περισσότερο αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ χωρίς μικρόφωνο. Θα σας ζητήσω τώρα, Επίτροπε, να απαντήσετε στις τελευταίες ερωτήσεις και να εξηγήσω και πάλι, κύριε Μπουτικόφερ, γιατί ήμουν... Ε, γιατί ε, δεν το περίμενα από πλευρά σα. Θα έπρεπε να είχατε ζητήσει από τον συνάδελφό σα, τον κύριο Γιάβορ, να σα δώσει το χρόνο των τριών λεπτών του και να ε, μπορέσετε έτσι να θέσετε όλα τα ερωτήματα. Κοιτάξτε. Ο, ο κύριος Μπουτικόφερ διακόπτη. Είναι άδικο αυτό που λέτε. Ναι, εσείς είστε άδικος, λέει ο κύριος Μπουτικόφερ. Μάλιστα. Κύριε Πίτροπο, έχετε το λόγο. Ναι, και έγινε λόγος για το copyright. Υπάρχουν αρμόδιες κατ' ουσίαν επιτροπές στο Κοινοβούλιο που έχουν λάβει το θέμα. Ε, πάντως, θα ήθελα εδώ να συνδέσω το ζήτημα του copyright γιατί η δημιουργική οικονομία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και στην πρόταση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του χρήστη για την πληροφορία, είτε είναι μουσική, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι ταινία οτιδήποτε είναι προσβάσιμο θα πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιεί, να το ακούει, να το βλέπει, να το διαβάζει και ταυτόχρονα προβλέπεται και μια αποζημίωση για τον ε, δημιουργικό κλάδο, είτε πρόκειται για τον σεναριογράφο, τον συγγραφέα, τον δημοσιογράφο, τον σκηνοθέτη, τον ε, συνθέτη, τον μουσικό, τον ε, τραγουδιστή ή τον ηθοποιό, καλύπτεται με μια δίκαιη αποζημίωση. Αυτός είναι... Αυτό είναι και το ζήτημα που μας γίνεται σε σχέση με, τον με την ποιοτική δημοσιογραφία. Στην ε, ε, Επιτροπή εδώ βιομηχανίας αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να συζητηθούν τα θέματα αυτά για τη δημιουργική οικονομία, αλλά αρμόδιες καθήλυν είναι άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Βέβαια πάντα είμαι στη θέση για περαιτέρω συζητήσεις. Ο κύριος Γαϊμόν ρώτησε ε, πώς προβλέπετε να γίνει αυτή η αλλαγή πόστου. Δεν έχω λάβει πρόταση από πλευράς της Βουλγαρίας για το ποιος ή ποια υποψήφιος υποψήφια θα εκπροσωπήσει την Βουλγαρία. Περιμένουμε την πρόταση. Ξέρετε ποια είναι και η πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Επομένως, το ποιος θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της, ευρω... της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, εάν έχει δηλαδή το προφίλ εκείνο ο υποψήφιος ή η υποψήφια που θα προταθεί από την Βουλγαρία για να λάβει αυτό το ε, χαρτοφυλάκιο, δεν το γνωρίζουμε. Είναι ένα ζήτημα ούτως ή άλλως το οποίο κρίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής αναλόγως με, την, ε, με, τις τα προσόντα, με το επαγγελματικό προφίλ κτλ. Άλλωστε έχει διορίσει και όλους τους, έχει κατανέμει τα χαρτοφυλάκια σε όλους τους ε, επιτρόπους. Εγώ πάντως έχω δεσμευθεί να παραμείνω μέχρι το Δεκέμβριο στη θέση αυτή και ενδεχομένως, αν χρειαστεί και μετά, να ε, λειτουργήσω ως σύμβουλος για τον διάδοχο στο θέμα της στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας. Για τον κύριο Μπόνι, που ρώτησε πώς ε, συμπεριφέρονται τα κράτη-μέλη στην υπόθεση. Εδώ έχουμε να κάνουμε διάφορους τομείς της πολιτικής που, ε, όπου σημειώνεται, όπου υπάρχει θέμα Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή διάσταση διαμόρφωση τη πολιτική, μια κάποια διστακτικότητα. Πάντω για το ψηφιακό τομέα μπορώ να πω ότι τα κράτη-μέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και στι επιμέρου ειδικέ ομάδε του Συμβουλίου γιατί χθε και σήμερα δύο φορέ ήμουν παρόν σε συνεδριά του Συμβουλίου ότι και είδα ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να δεχθούν τον εξευρωπαϊκισμό των κανόνων, των προτύπων, των προδιαγραφών και λοιπόν διατάξεων για τι αγορέ, διότι διαπιστώνουν ότι οι ψηφιακέ αγορέ δεν είναι ε, την ψηφιακή αγορά δεν μπορούν να διαμορφώσουν και να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστικότητα των Αμερικανών ή των Ασιατών ανταγωνιστών μας, τα κράτη μεμονωμένα. Για τον κύριο Μπιουτικόφερ και το Ράμι που πολύ εύστοχα ρώτησε. Ήμουνα στην ε, ετήσια συνάθρηση του IIC, βιομηχανία 4.0, στο Βάλντορφ, ε, προσκεκλημένος ως ομιλητής, κύριε Μπιτικόφερ, και θέλω να πω το εξής ότι λίγοι θα είναι οι τομεί όπου η βιομηχανία ενός κράτους μέλους στην Ευρώπη έχει προχωρήσει τόσο ώστε να έχει την παρακολούθηση των Bitcom και άλλων σημείων από ένα Υπουργείο. Ίσως η βιομηχανία 4.0 να μετατραπεί σε μια παγκόσμια εμβέλεια έννοια. Στην Αυστρία ήδη λέμε, λένε βιομηχανία 4.0 Αυστρίας. Ιταλία, στην Ιταλία λένε Ιταλίας. Εγώ ως Γερμανός βλέπω με χαρά ότι χρησιμοποιείται αυτή η έννοια, αλλά εγώ θα προτιμούσα να λέγαμε Digitalizing European Industry. Τώρα τι θα κάνει αυτή η πλατφόρμα ε, βιομηχανία 4.0 και αν θα αρκεί για ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτό είναι το κρίσιμο και γι' αυτό στο βαθμό του δυνατού ενσωματώνουμε την πλατφόρμα αυτή στην πλατφόρμα των πλατφορμών όπως την ονόμασα νωρίτερα που ιδρύσαμε πρόσφατα με εκπροσώπους από τη Smart Factory, του Βιομηχανία 4.0 και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα πλατφόρμα εκπροσωπούνται από ε, τις κυβερνήσεις τους. Πάντα κρίσιμο είναι το κράτος και είναι τώρα η Ρουμανία, η Ουγγαρία ή άλλο κράτος τώρα να μελετάει τη δυνατότητα ίδρυσης μιας εθνικής πλατφόρμας. Με τον κύριο Κούκα, Άικστρομ, Άρομ ή άλλη ε, επιχείρηση. Το ερώτημα πάντα είναι αν χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό δίκαιο εξωτερικών οικονομικών σχέσεων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Εγώ αυτό που κάνω το εξή. Είμαι αρμόδιος για 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν την έρευνα κάθε χρόνο ως Επίτροπος. 100 εκατομμύρια δίνουμε για τη ρομποτική παραδείγματι το χρόνο κύριε Κούκα. Και σας βεβαιώ ότι στον τομέα της έρευνας μπορούμε να δεχθούμε ως εταίρους μας μόνο εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, τόπο ερευνητικό, εγκαταστάσεις δηλαδή ερευνητικές και τεχνογνωσίας μέσα σε ευρωπαϊκό κράτος. Αυτή είναι η ΣΔΙΤ που έχουμε για τη ρομποτική, στο βαθμό που η εταιρεία αυτή έχει στο Augsburg τα εργαστήρια της ρομποτικής και που ε, παραμένει σε ευρωπαϊκή επικράτεια για την ανάπτυξη. Για την επόμενη λοιπόν δημοσιονομική περίοδο, για την περίοδο μετά το ορίζον 2020, που θα απασχολήσει το Κοινοβούλιο σας τα επόμενα δύο χρόνια ή σε δύο χρόνια καλύτερα, πάλι θα πρέπει να διαφυλαχθεί αυτή η αρχή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ενδιαφέροντος και ε, ε, έρευνα ανάπτυξη. Ανεξαρτήτως του ποιος διακρατά τις ε, μετοχές, πρέπει η έρευνα και η ανάπτυξη για την οποία είναι πολύ σημαντικές οι εταιρικέ αυτές σχέσεις εις ΔΙΤ, να παραμένουν στην Ευρώπη ε, ώστε να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή οικογένεια έρευνας και ανάπτυξης. Το άλλο θέμα μιας ε, κοινή νομοθεσίας για τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ρωτήσετε σε άλλο επίτροπο, άλλος θα πρέπει να απαντήσει. Εγώ πιστεύω πάντως όντως ότι θα πρέπει να υπάρχει, εφόσον υπάρχει ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και πρέπει να είναι αμφίδρομη η σχέση, δηλαδή εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και δεκτικοί όσο είναι ανοιχτέ και δεκτικές και οι λοιπές αγορές αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να σας απασχολήσει στο μέλλον ε, σε αυτό το χρόνο. Για την αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας και τον περιορισμό της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, τα smart cities και communities, ευφύς πόλεις και κοινότητες με συνεργασία της DigiHoof, της ε, Grow, της ε, Connect και της ENA έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη, σε συνεργασία με τις πόλεις εταίρους, πρότυπα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με περιορισμό των αναγκών σε μεταφορά με, με βελτιστοποίηση του τομέα των μεταφορών και με αποτελεσματικές ενεργειακές λύσεις για τα κτίρια σε ισότιμες λοιπόν συνθήκες διαβίωσης και βιομηχανικής παραγωγής θέλουμε οι ενεργειακοί όγκοι να περιορίζονται και βέβαια αντίστοιχα ιδιαίτερα να περιορίζονται οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Για τον κύριο Ρούμπιχ, για το χίδιν, ε, για, το, για, τη χίδιν, για, το, για περιαγωγή. Για τον επόμενο Ιούλιο έχουμε προβλέψει ήδη την κατάργηση των τελών περιαγωγής στις ευρωπαϊκές αγορές. Μέχρι το 2015 το Δεκέμβριο Είχαμε στην νομοθεσία Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα και το θέμα της ε, χίδιν περιαγωγής, του wholesale roaming και ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι και για το fair use, την ε, ε, ισότιμη χρήση. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε να συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τις προηγούμενες εβδομάδες ακούσαμε την Πέρι, τον κύκλο δηλαδή εκείνων των αρχών ρύθμισης. Υπάρχει επιτροπή, ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που ε, θα κρίνει την πρόταση και για το θέμα της ε, ισότιμης χρήσης υπάρχει ένα πρόβλημα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Λετωνία τα τέλη των ε, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι το ένα έκτο αυτών της Ιρλανδίας. Αν λοιπόν ένας Ιρλανδός πολίτης μετά την κατάρρευση της περιαγωγής, τον Ιούλιο του 2017, που πιστεύουμε ότι θα γίνει, αγοράσει μια κάρτα SIM ενός λετονού ε, παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χωρίς να είναι κάτοικος Λετωνίας αλλά ενωμένοι στο Δουβλίνο και χρησιμοποιεί τις τηλεπικοινωνίες μέσα στο Δουβλίνο για, τη, για τηλέφωνα ε, μέσα στην πόλη ή το Λονδίνο ή σε κάποια άλλη πόλη της, Αυστρία, της Ευρώπης τότε αυτός ο Λετωνός ε, πάροχος θα έχει ε, θα αγοράζει πιο ακριβά τις μονάδες μεταφορές αυτές της χίδη να πω ότι αν τις αγόραζε για χρήση στην εγχώρια αγορά. Αυτή η κατάχρηση εντός εισαγωγικών είναι στόχος μας να περιοριστεί χωρίς περιβολικές γραφειοκρατίες, χωρίς το όριο των 90 ημερών, χωρίς περιορισμό των ε, όγκων των μεταφερομένων δεδομένων, από ό,τι μας λένε οι δικοί μας, από ό,τι μας λένε και στην ομάδα εργασίας, αυτό, αυτή είναι η προσπάθεια στο Συμβούλιο, δηλαδή να δώσουμε μια λύση χωρίς αυτούς τους περιορισμούς. Πάντως, εάν αρχίσει να μπαίνει μέσα ο λετωνός πάροχος, τότε προφανώς και ο λετωνός εκπρόσωπος της κυβέρνησης ε, στην, ε, στο Συμβούλιο, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, θα ταχθεί κατά της πρότασης. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την κατάργηση και τήρηση των όρων κατάργησης του roaming τον Ιουλίο του 2017. Για το STE και το γνωρίζω καλά, ε, μπορώ να σας πω για τους ημιαγωγούς και τη, τη μικροηλεκτρονική, φέτος το Μάρτιο ξεκίνησα το πρόγραμμα εισαγωγών ε, για τις ευρωπαϊκές αγορές με 7 κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, οι κατοχώρες και δύο άλλες Αυστρία και Βέλγιο. είμαστε σε συνομιλίες λοιπόν μαζί τους και βέβαια και σε μια διάσκεψη συναντούμε τη βιομηχανία με εκπρόσωπο που μας ε, επένεσε διαιτέρως λέγοντας ότι με την εταιρική αυτή σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη, μέλη και βιομηχανία μπορούμε να τα καταφέρουμε τα μέσα, τα κονδύλια που μπόρεσα εγώ να εξασφαλίσω από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για τα πέντε κράτη-μέλη, μπορέσαμε να τα διπλασιάσουμε χάρη στην ε, συμβολή της βιομηχανίας και βέβαια πολλαπλασιαστικά και με τις ε, λοιπές προτάσεις. Πρέπει λοιπόν με δεδομένο τον ανταγωνισμό από τους Κινέζους και γενικά οι ε, ανταγωνιστές να έχουμε αυτή την πολλαπλασιαστική, αυτή τη μόχλευση. Η διάσκεψη αυτή της εβδομάδας στη Ρώμη ήταν πάρα πολύ καλή, επίσης ε, επιτυχημένη και είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης για την οδηγία ανής τώρα πρέπει αυτή να υλοποιηθεί στα κράτη-μέλη, δηλαδή να μεταγραφεί σε εθνικό δίκαιο και σκοπεύω ταχύτατα να προχωρήσω σε επικαιροποίηση γιατί η κυβερνοασφάλεια είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να κερδίσει, μπορεί, πάνω στο οποίο μπορεί να παιχθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη, στο cloud, στην ε, ε, βιομηχανική κατασκοπία, σε θέματα τρομοκρατίας. Έχει τεράστια σημασία η κυβερνοασφάλεια. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα θέμα που έχει να κάνει με ευρωπαϊκή ευρωπαϊκές νοοτροπίες, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Σας ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Uh, thank uh, ε, we Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σας ε, ξαναδούμε στο μέλλον, κύριε Επίτροπε, ως Αντιπρόεδρο για τον προπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, όπως έχει ανακοινωθεί ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη σπουδαία σας δουλειά. για την ψηφιακή οικονομία και για τον διαρκή διαρθρωμένο διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή Ήτρε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εσάς ως εκπρόσωπό της. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Έχουμε αργήσει αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, το επόμενο θέμα τώρα είναι οι εκπομπές ε, των αριών θερμοκηπίου και την συμπέριληψή του ε, και την απορροφή από τη χρήση γη, τι αλλαγέ στη χρήση γη και τη δασοκομεία στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια μέσω του 2030. Η Μαρίζα Ματία είναι η εισηγήτρια από την ΚΟΕ. Θέλω να σα θυμίσω ότι οι εκπομπέ και η συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γη και τι αλλαγέ στη χρήση γη και τα νοσοκομεία καλύπτονται μόνο από τι διεθνεί μα υποχρεώσει στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιώτο και τίποτε άλλο. Το πρωτόκολλο του Κιώτο ε, αναφέρει μια σειρά από ε, περιορισμούς στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της, έτσι ώστε η αλλαγή χρήσης γης και ε, η στρατηγική για τη δασοκομεία ε, να μην δημιουργούν περαιτέρω εκπομπές. Ο στόχος πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια πρόταση της οποίας το αντικείμενο είναι να καθορίσουμε πώς θα συμπεριλάβουμε αυτό το κλάδο στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 και μετά θα υπάρξει γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε προς την Επιτροπή Ένβη που είναι η βασική επιτροπή για το θέμα αυτό. Μια σειρά από πτυχές που έχουν να κάνουν με τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τη δασοκομεία ε, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Επιτροπή μας. Παραδείγματος χάρη επιπτώσεις της, της αλλαγής χρήσης γης για την ε, γεωργία, την δασοκομική βιομάζα για ενεργειακή χρήση, αλλά και ε, άλλων πρώτων υλών για τη βιομηχανία μας. Πολλά λοιπόν ζητήματα. Η συνάδελφος Μαρίσα Ματίας ε, παρακαλώ να ανοίξει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε, γιατί ήδη έτσι με ξαλαφρώνει από ένα μεγάλο κομμάτι της δικής μου εισήγησης. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε σε σχέση με αυτή την έκθεση. Είναι ένα σημαντικό ε, θέμα και γι' αυτό πιστεύω πως η πρόταση της Κομισιόν είναι ευπρόσδεκτη, όπως, ε, καθώς αναφέρεται σε αυτά τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλου του Κιώτο και είναι περιορισμένη η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να μπορέσουμε μετά το 2020 και ε, να, αντιδράσουμε και κυρίως χρειαζόμαστε αποφάσεις ώστε να λάβουμε υπόψη την επίτευξη των όσων συμφωνήθηκαν στο Παρίσι σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύω ότι βεβαίως ε, δεν είμαστε εμεί αρμόδιοι από τη Επιτροπή, αλλά έχουμε εδώ ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στη γνωμοδότησή μας. Σήμερα θα ακούσουμε και τους κοιόδης εισηγητές και θα καταλάβουμε λίγο ποιες είναι οι απόψεις τους, αλλά Α, όσον πρόκειται για την αλλαγή, τη χρήση γης, την αλλαγή χρήση γης και τα δάση, υπάρχουν διαστάσεις όσον αφορά τις εκπομπές, διαστάσεις που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Θα ήθελα εξ αρχή να σας αποσαφηνίσω ότι συμφωνώ με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ελπίζω ότι θα διατηρηθεί ε, η άποψη αυτή στη διάρκεια τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ λοιπόν με την προσέγγιση για τη χρήση γη την αλλαγή χρήση γης και τη δασοπονία πέρα από άλλα συστήματα και προγράμματα που ήδη υπάρχουν, ε, δηλαδή όταν μιλάμε για παράδειγμα για το σύστημα Εμπορία εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών το ETS, γιατί νομίζω πως πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση και πρέπει να το συζητήσουμε και ξεχωριστά. Ω προ αυτό και όσον αφορά τη δική μας Επιτροπή, πιστεύω θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, τη βιομηχανία και τι μεταφορέ. Καθώς επίσης να λάβουμε υπόψη πω οι αλλαγέ που γίνονται σε σχέση με την οικονομία που εξαρτάται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα δεν θα αμφισβητήσει τα μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν για τον περιορισμό των εκπομπών στην περίπτωση της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και των δασών. Κάτι ακόμα που ίσως να μην έχει απόλυτη σχέση με την Επιτροπή μα, ωστόσο πιστεύω θα πρέπει να το λάβουμε επίση υπόψη, είναι το να επικεντρώσουμε όλη αυτή την προοπτική μέσα σε μια γραμμή προσέγγισης που ευνοεί την βιοπικιλότητα, την ποιότητα του, της γης, την ποιότητα του νερού Εν πάση περιπτώσει, ζητήματα που δεν έχουν άμεσα ε, σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, αλλά με την ε, έρευνα και την καινοτομία. Άρα λοιπόν πέρα από τον τομέα των μεταφορών της τεχνολογίας και της βιομηχανίας πιστεύω ότι η έρευνα και η καινοτομία εδώ είναι απαραίτητες και θεμελιώδεις και από αυτή την άποψη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ζητήματα της βιοπικιλότητας και τα όσα ήδη ανέφερα. Τρίτη μου παρατήρηση. και αυτό διέπει την γνώμη μου για όλες τις επιτροπές ε, και η δική μας εδώ δεν αποτελεί εξαίρεση, είναι το θέμα της διαφάνειας και στους τομείς που ε, μας απασχολούν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στα ζητήματα διαφάνειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πηγές των δεδομένων, τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ε, για να έχουμε ευκόλυνση στα συστήματα ενημέρωσης, αλλά να έχουμε και συγκρίσιμες και εξολογήσιμες πληροφορίες που θα συλλέγονται με ισότιμο και διαφανή τρόπο στο πλαίσιο των, από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, δεν θέλω βέβαια να επεμείνω στα δικά μου. Θέλω να ακούσω τα όσα έχουν να οι συνάδελφοι από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, ώστε να έχω μια πιο ε, ολοκληρωμένη εικόνα στη, κατά τη σύνταξη του σχεδίου γνωμοδότησης, αλλά και πάλι, όπως είπα, ό,τι έχει να κάνει με τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις μεταφορές και το θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης, που είναι, κατά τη γνώμη μου, οι προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιούσο, εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την παρέμβασή της. Πρόκειται για μια πρώτη συζήτηση. Εγώ θα αναφερθώ απλώς σε κάποιες ανησυχίες ε, που με απασχολούν. Πρώτα απ' όλα αυτή η πρόταση ε, σχετίζεται άμεσα με αυτή που έχει να κάνει ε, με τους τομείς που περιλαμβάνονται στο σύστημα ανταλλαγής ε, εκπομπών. Ε, αυτοί που δεν περιλαμβάνονται και βεβαίως αυτοί που έχουν να κάνουν με την ε, κατανομή του, της προσπάθειας από τα κράτη-μέλη. Ε, θέλουμε εδώ να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν παράλληλα να εξετάσουν οι προτάσεις. Δεν μου φαίνεται κακό να τα δούμε ταυτόχρονα, διότι είναι κάτι που συνδέεται και με την πρόταση για το, την εμπορία ε, εκπομπών και των τομέων που εμπλέκονται, που εντάσσονται στο σύστημα αυτό. Υπάρχουν δύο περίοδοι ε, στην πρόταση αυτή, 2021 έως 2025, η πρώτη. Στις περίοδους αυτές ε, μπορούμε να έχουμε μέρος της απορρόφησης εκπομπών από τη μία χώρα στην άλλη ή από τη μία περίοδο προς την άλλη. Η ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι η εξή. Μετά την τελευταία περίοδο, 2026-2030 δηλαδή, εάν υπάρχει πλεόνασμα απορροφήσεων, μπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη περίοδο ή σε άλλο κράτος μέλος, είναι ένα ερώτημα που ήθελα να υποβάλω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα προϊόντα ξυλίας, τα επεξεργασμένα. Ε, καλό ακούγεται αυτό. Βεβαίως είναι περίπλοκη η μαθηματική φόρμουλα. Η συγγήτρια αναφέρθηκε στη διαφάνεια. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω είναι να υπάρχουν κανόνες που να είναι ομοιογενείς για όλα τα κράτη-μέλη. Διότι σε αυτή τη φόρμουλα που μας υποβάλλεται, που μας παρουσιάζεται, με την, ε, τον κύκλο ζωής του ξύλου και, και τις διάφορες, ε, τα υπόλοιπα ξυλίας που πάνε στα, στα απόβλητα, είναι μικρές, ε, μικρές οι διακυμάνσεις. Να κάνω άλλο ένα ερώτημα αυτό το όριο των 280 εκατομμυρίων τόνων που έχει θέσει η Κομισιόν ε, θα μπορούσε να αυξηθεί. Ένα ακόμα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Κομπούλα Νάτρη τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είπε η συγκήτρια ότι αυτά που είναι σημαντικά για την Επιτροπή Ήτρε ε, θα αποσταλούν στην, ε, και στην ένβη που θα έχει αυτή η άποψη. Όταν μιλάμε όμως πάντα για τα δάση, μιλάμε για τόσα ζητήματα, όταν μιλάμε για τη γεωργία πάλι καλύπτουμε, αυτό αγγίζει πολλούς τομείς, είναι αδύνατο να μιλήσουμε για τις καινοτομίες ε, για το μέλλον, για την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να λάβουμε υπόψη μας και τη βιοοικονομία. Έτσι λοιπόν η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά καλή ως βάση θα πρέπει να απαντήσουμε, να αντιδράσουμε στην ε, κλιματική αλλαγή και βεβαίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως δεξαμενή αυτά τα στοιχεία, αλλά ακόμα και μια δεξαμενή έχει τα όριά της, είναι καλύτερο ε, να είναι βιώσιμος, ε, βιώσιμη αυτή η δεξαμενή και αυτό το έχει πει και αυτή η Επιτροπή για τη, δασοκομία, για τη στρατική δασοκομεία. στο να έχουμε μια καλύτερη, να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη δασοκομεία, τότε θα έχουμε περισσότερες ίνες. Ε, και αυτό μπορεί να βοηθήσει για να παράγουμε καινοτόμα βιολογικά προϊόντα και να βρούμε νέους τρόπους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή μας να κοιτάξει προς το μέλλον. Η πρόταση της Κομισιόν κοιτάζει προς τα πίσω, κοιτάζει στα έτη 90-2009. αλλά Θα πρέπει να πάμε προς τα μπρος, να δούμε ποια είναι τα κίνητρα για να μπορέσουμε να φροντίσουμε καλύτερα τη γη μας. Ε, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί είναι εξαιρετικά σοβαροί και νωρίτερα μιλήσαμε για την ευελιξία η χρήση υγιής, τα ETS είναι μέρος της ευελιξίας αυτής και αυτοί οι στόχοι βεβαίως που έχουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τη συνολική εικόνα. Αλλά το βασικό κίνητρο για μένα σε αυτήν την έκθεση είναι να δοθούν κίνητρα ε, για την ε, παραγωγή ξυλίας που να λαμβάνει υπόψη τις πρώτες ύλες, ε, τις δεξαμενές, τη διατροφή, όλα αυτά τα αισθήματα τα, τα οποία μπορεί να συνεισφέρει τα νοσοκομεία. Αυτά ευχαριστώ. Από την Άλντε τώρα ο συνάδελφος Φέντερλεϊ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια ε, για τις αρχικές σας ε, παρατηρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ε, για να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην δημιουργήσουμε νομοθεσία που θα εμποδίσει την οικονομία, θα θέσει πραγμού στην οικονομία, όπως είπε και η κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Γνωρίζουμε πολύ λίγα σήμερα για το τι μπορεί να παράγει πράγματι το δάσος. Γι' αυτό θα ήθελα να δω και και κάποιες αναφορές σε υποκατάσταση, γιατί υπάρχει μια αγορά όπου χημικά που σήμερα γίνονται με βάση συστατικά ε, ορυκτά, από, τα, από ορυκτά, ε, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν υποκατάστατα από, από τα δάση. Ας πούμε τα υφάσματα πολύ συχνά ε, κατασκευάζονται από σελουλόζη. που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και χρησιμοποιεί λιγότερο νερό ε, για την παραγωγή βάμβακος, ε, μακερών μάλλον υφασμάτων. Επίσης είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για τις θέσεις απασχόλησης στις περιοχές της υπαίθρου ε, και συμβάλλουν σε κάποιες χώρες πολύ στην οικονομία της χώρας. Φιλανδία, Σουηδία, Αυστρία είναι με χώρες όπου η δασοκομεία συμβάλλει σε τεράστιο ποσοστό. Ας πούμε, πέρυσι η δασοκομεία παρέγει τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι η Σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία. Uh, uh, το να διατηρηθούν ε, τα, οι αποθήκες άνθρακα ενώ χρησιμοποιούν, χρησιμοποιείται ενέργεια ε, από τα δάση μπορεί να οδηγήσει στα καλύτερα ωφέλη όσον αφορά την μετρίαση, τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αλλαγών. Χρειάζεται ένα σύνολο κανόνων που θα είναι εύκολο να υπολογιστούν και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι το γεγονός ότι η διαχείριση των δασών γίνεται με διαφορετικό τρόπο και έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε εμπόδια στους υπολογισμούς ε, αυτούς. Για σε ορισμένα μέρη της, Ελλάδα, ε, της Ευρώπης γίνεται προσπάθεια για αναδάσωση ε, σε νησιά, ας πούμε, ενώ στη Σουηδία, τη Φιλανδία, εδώ και 150-200 χρόνια έχουμε έναν αναπτυσσόμενο τομέα του ξύλου. Στις χώρες όλες αναπτύσσεται ο τομέας της δασοκομείας, αλλά βλέπουμε ότι σε άλλες Χώρε χώρες είναι τεράστιο πρόβλημα η ε, αποψήλωση των δασών και πρέπει να αλλάχθούν υπόψη οι διαφορές αυτές. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής εξ των Πρασίνων, ο κύριος Γιάβορ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία της. Έχουμε, καλωσορίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για την ενεργειακή πολιτική. Εν γέννη, ε, βλέπουμε θετικά την πρόταση της Κομισιόν, ωστόσο υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτίωση. Σύντομα να αναφέρω τρεις πτυχές του κανονισμού όπου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας κατά τη γραμμή. Πρώτον, επίπεδο φιλοδοξίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συμβάλλει ο τομέας αυτός στην επίτευξη των στόχων ε, που ανέλαβε, των δεσμεύσεων μάλλον της Ένωσης υπό τη Συμφωνία του Παρισιού, τριασμό των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των δασών ως πηγής αρνητικών εκπομπών. Αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να αποτελέσει ένα εργαλείο για να ε, προωθηθεί ο ρόλο των δασών ώστε να μπορούν να αποθηκεύουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να περιορίσουμε τη θέρμανση κάτω από τον 1,5 Βαθμό. Ε, δεύτερον, ε, κανόνες λογιστικής καταγραφής. Αν και η Κομισιόν ε, βελτιώνει του κανόνε καταγραφή, ε, εξακολουθεί να προτείνει τρει διαφορετικέ μεθόδου λογιστική καταγραφή, πράγμα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαφάνεια του συστήματο και να επιτρέψει παραθυράκια. Τρίτον, βιώσιμη χρήση βιομάζας. Πάλι είναι πολύ σημαντικό ότι η LULUCF, δηλαδή η χρήση γης, αλλαγής χρήση γης και η δασοπονία, χρησιμοποιούν ε, διαφορετικούς τρόπους, δεν αυξάνει την αποθήκευση στο, στόκα άνθρακα, ε, γιατί μόνο βιώσιμη διαχείριση μπορεί να παράγει βιοκαύσιμα. Εν κατακλείδη να πω ότι αυτό, η χρήση γης, η αλλαγή χρήση γη και δεσοπονία είναι πολύ κρίσιμο πυλώνας μαζί με το ETS και το κανονισμό για την κοινή ε, προσπάθεια. Γι' αυτό και προσβλέπω στη στενή συνεργασία με τους συναδέλφους της ΣΥΤΡΕ και την εισηγήτρια και τους κοιόδης ώστε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την πρόταση Λουλού CF της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος για τις παρατηρήσεις σας και εξ ονόματος της ΓΚΟΕ έχουμε τον κύριο Κόχλιτσεκ, τον Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω αρκετές πρακτικού τύπου παρατηρήσεις. Βεβαίως, ο υπολογισμός των ωφελών όσον αφορά την ε, συλλογή τη σύλληψη, άνθρακα είναι πολύ σημαντική, ε, σημαντικός. Όμως ε, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στη Σουηδία ή στην Νότια Ιταλία ή στην Ισπανία. Το μόνο που μπορώ να συστήσω είναι να, γίνει ένας υπολογισμός, να γίνεται ένας υπολογισμός γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε διαφορετικού τύπου, γιατί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον ίδιο τρόπο στο βορρά και στο νότο. Πριν από 30 χρόνια περίπου έγιναν προσπάθειες για βελτίωση της ισορροπίας του διοξιδίου του άνθρακα μέσω της αναδάσωσης ε, και εκτός Ευρώπης. Για παράδειγμα, στην Αλγερία έγινε ένα τεράστιο πρόγραμμα για αναδάσωση του, του βόρειου άκρου της Σαχάρα. πράγμα που θα έχει επιρροή και στο Μαρόκο και Επίσης στην, στο νότιο άκρο της ε, ρήμου Γκόμπι οι Κινέζοι προσπάθησαν να αναδασώσουν ε, γιατί αυτό θα έχει μεγάλες, ε, μεγάλη επιρροή στις μεγάλες πόλεις όπως στο Πεκίνο. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό αυτά τα project αναδάσωσης που έγιναν, όπως είπα, σε πολλά μέρη του κόσμου θα πρέπει εδώ να συμπεριληφθούν Και άλλο ένα σχόλιο, 70% του πλανήτη είναι ωκεανοί. Στα μέσα του Ατλαντικού υπάρχουν τεράστια κομμάτια, τεράστια όγκοι πλαστικού. φαίνεται σαν ότι έχουν σχηματιστεί παγετώνες πλαστικού. Ε, δηλαδή είναι έρημη θάλασσα, είναι το αποτέλεσμα των απορριμμάτων που ρίπτονται στη θάλασσα μέσω των ποταμών. Αυτό το πλαστικό μολύνει και ρηπαίνει παντού, είτε πλέει στην επιφάνεια του ωκεανού, ε, και από ό,τι φαίνεται η αυτό το, το, ο όγκο πλαστικού είναι μεγαλύτερο από ολόκληρη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σκεφτούμε ριζικέ λύσει. Είναι τεράστιο κίνδυνο για τον πλανήτη μα και πραγματικό κίνδυνο. Αυτά λοιπόν τα πλαστικά νησιά σημαίνει ότι οι, οι, ακτίδες του ήλιου δεν μπορούν να τα διαπεράσουν και άρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί ζωή εκεί. Ο κύριος Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής με τα γενικά σχόλια που διατυπώθηκαν και με... Ε, να σας πω ότι εκπροσώπησα το Κοινοβούλιο στο Μαρακές στην κοπα 22. Ήταν εθαρρυντικό ότι τώρα θα αρχίσουμε την εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλάβουμε στο Παρίσι. Και το μήνυμα είναι ότι κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητα έχει ρόλο να παίξει και καμία περιοχή, κανένα τομέα δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Και φυσικά τα δάση έχουν τεράστιο ρόλο να παίξουν τόσο όσον αφορά το μετριασμό των εκπομπών, την μείωση των εκπομπών, όσο και την ενεργή, ενέργεια μέσω της βιομάζα, βιομάζας. Αρκετοί συναδελφοί τόνισαν ότι ο υπολογισμό και η λογιστική καταγραφή είναι πολύ σημαντικά, Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα για ενέργεια από την βιομάζα. Υπάρχει μια τάση να λέμε ότι ναι, υπέροχο είναι ανανεώσιμη κτλ. Όμως έχει υπολογιστεί ολόκληρη οικονομική δραστηριότητα από την καλλιέργεια στη μεταφορά κτλ. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε νομίζω. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε τα δάση όσον αφορά την κυκλική οικονομία. Το να έχουμε μια φυσική και παραγωγική ζωή μέχρι την τελική χρήση. Και είναι πολύ λογικό ότι ο κόσμος καλωσορίζει τις σύνες και τα λοιπά. Και αυτό πρέπει να το εθαρρύνουμε. Τελευταία μου παρατήρηση, και αυτό βέβαια συνδέεται με την κοινή γεωρική πολιτική και την μεταρρύθμιση της Εκεί θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να αναδασώσει. Ιδιαίτερα σε περιοχές περιθωριακές που τώρα χρησιμοποιούνται σχεδόν για μη κερδοσκοπικές εταιρείες ε, παραγωγής βόλου ε, κρέατος που αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί και να γίνει και πιο επικερδές μέσω της δασοκοπονίας. Πολλά πρέπει να γίνουν και αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φανχάιν, Τριματάρχης, Χρήση Γης, Καινοτομία, Γενική Επιτροπή για το Κλίμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να δώσουμε σύντομες απαντήσεις εκ μέρους Ευρωπαϊκής Χαίρομαι ιδιαίτερως που η Επιτροπή σας εξετάζει το θέμα αυτό σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. Η χρήση γης, η αλλαγή χρήσης και η ε, δασοκομεία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να πω ότι δεν είναι καινούργιο το θέμα. Έχει ήδη ρυθμιστεί υπό το πρωτόκολλο του Κιώτο και έχουμε και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καλύτερα απόφαση του 2013, που ήδη έχει σημειώσει τα πρώτα της βήματα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Κλίμα. Ιδιαίτερα λοιπόν είχαμε να κάνουμε τους κανόνες παρακολούθησης και καταγραφής, ώστε να έχουμε τις ε, γνώσεις για το τι σήμαινε η κάθε δραστηριότητα. Πρόοδο έχουμε σημειώσει και η νέα μας, πρόοδος, ε, η μας έκθεση, πρόταση τώρα βασίζεται πάντα στο πρωτόκολλο του Κιώτο και το εγγράφει στην, ε, στους στόχους για, την, για το κλίμα και την ενέργεια του 2013. Και εσύ θα, θέλαμε και αυτός το τομέας. Λουλουευσή να προχωρήσει έτσι ώστε να μην παράγει επιπλέον εκπομπές. Για το μέλλον. Ενθαρρύνουμε ενεργό διαχείριση των δασών ως μέσο χρήσιμο και θετικό και για το κλίμα, γιατί μπορεί να βελτιώσει και την παραγωγή ξύλου που υποκαθιστά υλικό ορυκτής προέλευσης και για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί για τα προϊόντα ξυλίας που επίσης περιλαμβάνονται και στην δική μας πρόταση γιατί μπορεί να έχουν πολύ θετική ε, απήχηση και καλύπτουμε με τις προτάσεις μας την δότα χρήση και, χρήσης και υπολογισμού ώστε να καταγράφεται ο αριθμός των ε, αφαιρέσεων εν πρόκειται για ξυλοεία, οικοδομών, πώς μπορεί να ενισχύσει την υφιστάμενη, τους εκτό υπολογισμούς εκτός ατμόσφαιρας. Γενικά τα προϊόντα της ξυλίας έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο ε, ποσοστού υποκατάστασης. Οι δεσμοί επίσης μεταξύ της πρόταση για τη χρήση γης και το εις πρόταση κανονισμού για τους τομείς ε, εκτός ETS επιτρέπουν μια ευελιξία. 280 εκατομμύρια τόνοι. Προσπάθεια που καλύπτεται και στη σχετική μελέτη επιπτώσεων. Μια τρίτη ε, ερώτηση είχε να κάνει με την καταμέτρηση ξυλίας για διαχείριση δασών, όπου πάλι πιστεύω έχουμε μια μοναδική προσέγγιση, γιατί προτείνουμε στα κράτη-μέλη να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία αναφορά. με επαλήθευση κάθε φορά της προσέγγισης ως το 2020. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι θετικά, διότι επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ε, λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ε, των δασών τους ε, κάθε φορά. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που έχουμε μέχρι τώρα λάβει και βεβαίως προσβλέπουμε σε περαιτέρω καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέγει ο Πρόεδρος, για τις παρατηρήσεις εκ μέρους Γενικής Διεύθυνση για το κλίμα και το λόγο θα λάβει η κυρία Ματίας, αν θέλει να πει δύο λόγια για το τέλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, στην ε, εισήγησή μου, όπως είπα, δεν έφυξα όλα τα ζητήματα ε, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτού του θέματος, αλλά βεβαίως υπάρχουν και περιορισμοί στην εκπόνηση μιας νομοδότησης, ιδιαίτερα σε μια, στο πλαίσιο μιας επιτροπής ε, συμβουλευτικής. Ωστόσο, αναφέρθηκαν ζητήματα που θα τα, λάβω υπόψη, γιατί είναι πολύ σημαντικά. κάναμε ε, έναν γύρο για θέματα ε, κινήτρων, για θέματα μετριασμού. Πιστεύω πως όλες οι παρεμβάσεις ε, ήταν ενδιαφέρουσες για να μπορέσω να συντάξω αυτό το σχέδιο, αλλά βεβαίως μεγάλο κομμάτι της δουλειάς θα γίνει μετά από την υποβολή του σχεδίου γνωμοδοτησής μου και το θα έχουμε την ευκαιρία να συμπληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ όλους. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρονοδιάγραμμα. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης 22 και 23 Μαρτίου. Η προθεσμία υποβολή τροπολογιών και ψηφοφορία εδώ στις 11 Μαΐου και ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ 22 Ιουνίου. Ψηφοφορία δε στην Ολομέλεια. Θα δούμε, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο τελευταίο σημείο για απόψε. Αποστολή Ήτρε στην Πορτογαλία και την Ισπανία. 2 με 4 Νοεμβρίου 2016. Ενημέρωση. Και αντιπροσωπεία που έπρεπε να μάθει τις δυσκολίες αλλά και τις επιτυχίες δύο νοτίων περιφερειακών χωρών. Γιατί, δεν ξέρω γιατί είναι περιφερειακές. τη γνώμη είναι στην καρδιά της Ευρώπης οι δυο αυτές χώρες. Μάλλον κάποια παρεξήγηση έχει γίνει εδώ. Ε, συμμετοχή στο Horizon 2020 και εφαρμογή της ενδιάμεσης έκθεσης. Επειδή εκπροσωπεί την καρδιά της Ευρώπης λοιπόν η κυρία Καμπεσόν Ρουΐς που είναι μέλος της Επιτροπής μας από τους σοσιαλιστές αλλά αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ίδρυ, ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπής αυτής και θα μας πει όλα όσα θέλει να μας πει για την επίσκεψη αυτή που ήταν πολύ σημαντική για την Επιτροπή Ήτρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, διερμηνείς μας να καθίσουν ακόμα. Α, όχι, εντάξει, έχουμε χρόνο, είμαστε ok. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε αυτές οι περιφερειακές χώρες, οι νότιες χώρες να βρεθούν όντω στην καρδιά του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ο στόχος της αποστολής αυτής στην Πορτογαλία και στην Ισπανία ήταν να μελετήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες με μικρότερη, μικρότερα ποσοστά συμμετοχή από το ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα έρευνας όπως ε, το Όριζας 2020. Θέλαμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες, ε, να δούμε τις διάφορες προτάσεις ε, που θα μας έκαναν την πρώτη μέρα 2 Νοεμβρίου ήμασταν στη Λισαβόνα συναντηθήκαμε με με το Ίδρυμα για την Επιστήμη και Τεχνολογία καθώς και με το Επιμελητήριο Έρευνας και εκπροσώπους ερευνητών στον τομέα της ενέργειας, του ύδατος, της γεωργίας ε, ή της ε, ανθρώπινες και κοινωνικές επιστήμες. Μεταξύ των βασικών μηνυμάτων που μας έδωσαν οι αρχές, οι τοπικές καθώς και εκπρόσωποι του τομέα της έρευνας στην Πορτογαλία ε, ήταν η δυσκολία του να αποτελέσει κάποιος μέρος ενός συγκεκριμένου PPP έγινε αναφορά στην δικασία συμμετοχή στο Ίμι και υπόθηκε επίσης ότι πρέπει να είναι πιο μικρές οι δράσεις. Δίνεται η εντύπωση ότι αυτά τα PPP ουσιαστικά αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις πολυεθνικές και αυτό δυσκολεύει τη συμμετοχή μικρότερων οργανισμών όπως αυτούς με τους οποίους συζητήσαμε. Επίσης, ε, ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της, ε, των επιδοτήσεων. Υπάρχει τάση οι, οι επιδοτήσεις να καθιστούνται από, από δάνεια. Βεβαίως, ε, ανάλογα με την κάθε οντότητα ταιριάζει διαφορετικός τρόπος χρηματοδότησης και πρέπει να μελετάτε αυτό πριν ε, να καταργούμε αυτόματα τις επιδοτήσεις προς όφελος των ε, δανείων. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της πρότασης, πέρα από τη διαφάνεια, αυτό που ζητούν είναι η αξιολόγηση ε, να είναι ποιοτική, να είναι ακριβής και βεβαίως να σχετίζεται με το αντικείμενο αξιολόγησης. Ε, ζήτησαν δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης και να υπάρχει το κατάλληλο, το κατάλληλο feedback όταν λαμβάνει η χώρα η, αξιολόγηση των διαφόρων project. Επίσης, αναφέρθηκε η ανάγκη να δοθούν μεγαλύτερε ευκαιρίε για τι ανθρώπινε και κοινωνικέ επιστήμε ε, στου πυλώνε 2 και 3 του κοινωνικού κλάδου και επίση θα πρέπει να διευκρινιστεί η ε, διεπιστημονικότητα των διαφόρων ε, δράσεων. Στο επόμενο πρόγραμμα, στο 1 τόμα, ζητήθηκε οι ανθρώπινε και κοινωνικέ επιστήμε να έχουν πιο σημαντικό ρόλο από την οριζόντα 2020 γίνεται αναφορά στον όριο του 2020 στις επιστήμες, αλλά δεν εξετάζεται η, ε, να μην εξετάζεται μόνο η, η απόδοση οικονομική σε βραχυπρόθεσμο στάδιο. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τώρα, για αναφορά στους εξωτερικούς οργανισμούς, ε, και με τι Ισπανικέ Αρχέ υπόθηκε αυτό. Δεν υπάρχει επαρκή συγχρονισμό των διαστροτικών ταμείων, επαρκή συντονισμό ε, και με άλλα ταμεία. Στα πλαίσια του Οριζόντα 2020 έγινε αναφορά επίση ε, στην νομοθεσία περικρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζεται ε, στα διαστροτικά ταμεία που καθιστά αδύνατη τη συμβατότητα μεταξύ των δύο νομοθεσιών, δηλαδή αυτή των διαστροτικών ταμείων με αυτή του Οριζόντα 2020. Επίσης ζητήθηκε να εστιάσουμε περισσότερο σε μια δράση, σε δράση από κάτω προς τα πάνω, στα πλαίσια του 2020, για να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Επίσης υπόθηκε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι τομείς στον 2020 που αφορούν την απόδοση ε, του, ε, της έρευνας και εκεί η περιφερειακέ χώρε θα μπορούσαν να παίξουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Τη δεύτερη μέρα ήμασταν στην Ισπανία, στο Κάντιθ πιο συγκεκριμένα, στην έδρα του Διεθνού Κάμπου Αριστεία των Επιστημών τη Θάλασσα, με ε, τον αντιπρίτανη τη περιοχή τη Ανταλουσία, της Πανεπιστημίου της Ανταλουσία μάλλον, ε, υπάρχουν 14 κέντρα έρευνα που συμμετέχουν ε, εκεί που προέρχονται από τρεις χώρες, ε, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο και συντονίζει το Πανεπιστημίο του Κάντιθ. Έχουμε να κάνουμε εδώ με την γαλάζια ανάπτυξη το 2020. 17 spin-off ε, έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή από αυτό το σχήμα. Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να χρηματοδοτήσει ΣΔΙΤ για την γαλάζια ανάπτυξη η, η γαλάζια οικονομία και η γαλάζια ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει μια πραγματική κοινωνική πρόκληση για το επόμενο πρόγραμμα, το ένατο. Επίση, έγινε αναφορά στο γεγονό ότι οι χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσει, ε, πολλέ μικρέ επιχειρήσει και είναι σημαντικό να υπάρχουν ενδιάμεσα προγράμματα και projects τα οποία να μπορούν να συμμετάσχουν. Ένα άλλο θέμα που επανήλθε και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία είναι το χάσμα που υπάρχει ε, μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλά, υψηλές οι απαιτήσει και τα κριτήρια για τις, μικρομεσαίες, για τις ε, επιχειρήσεις και ότι πρέπει τα συγκεκριμένα κριτήρια να προσαρμοστούν. Την τελευταία μέρα, την τέταρτη μέρα στην Ανδαλουσία, συναντήσαμε του εκπροσώπου τη κυβέρνηση τη Ανδαλουσία καθώ και του εκπροσώπου του Τεχνολογικού Κέντρου για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη τη Ισπανία και το Ανώτατο Συμβούλιο Έρευνας μας είπαν και αυτοί τις απόψεις τους. Πρέπει εδώ να ξεχωρίσουμε ε, αυτά που μας είπε η κυβέρνηση της Ανταλουσίας ε, αλλά και η πορτογαλική κυβέρνηση αναφέρθηκαν στην στην αρχή της προσθετικότητας που δεν είναι η κατάλληλη σε ό,τι αφορά τα θεωρητικά ταμεία. Δηλαδή η κυβέρνηση υποκαθιστά τα, τα, τα κονδύλια έρευνα των διαφορετικών ταμείων και έτσι δεν λαμβάνεται υπόψη την αρχή της προσθετικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα των διαφορετικών ταμείων και αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ζητήθηκε λοιπόν να υπάρξει κάποια τροποποίηση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε ε, να μπορεί ένα κράτος μέλος ε, να έχει το περιθώριο λιγμών αλλά να μπορεί να γίνουν εν μεταφορές από, την, από το ένα project στο άλλο. Πρέπει να πούμε ότι πάει καλά στην Ισπανία η συμμετοχή στο σύστημα, το μεγάλο, στο, πρόγραμμα μάλλον, τα προβλήματα που αναφέρθηκαν για την Ισπανία είναι πανεφέρει με αυτά της Πορτογαλίας, υπάρχει, υπάρχει υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής και είναι λιγότερα τα προβλήματα. Ένα βασικό σημείο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ισπανία είναι ότι υπάρχει μια δομή και μια υποστήριξη από το ίδιο κέντρο, το τεχνολογικό, τεχνολογικό κέντρο βιομηχανικής ανάπτυξης που είναι ένας ε, δημόσιος φορέας που παίζει ένα ρόλο συντονισμού εξαιρετικά σημαντικό και έτσι η συμμετοχή της Ισπανίας στον 2020 είναι σημαντική ε, και σε αυτό το πρόγραμμα και στο προηγούμενο. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ζωρίνιο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν συμμετείχα στην επίσημη αποστολή, αλλά επειδή ως μέλος της Ήτρε και ευρωβουλευτής που εκλέγομαι σε αυτή την ε, κεντρική χώρα της Ευρώπης που είναι η Πορτογαλία Παρακολούθησα τις ε, ελέγχους που έγιναν στη χώρα μου. Ήταν πολύ σημαντική έλεγχη που μας ε, βοήθησε να δούμε ακριβώς που βρίσκεται η κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η συνάδελφος ε, Καμπεθόν Ρουίς ήδη μίλησε πληρέστατα για το τι συμβαίνει και ανέλησε και τις ιδέες της ε, εγώ θέλω να μιλήσω για τη διεύρυνση του φάσματος χρηματοδότησης για πιο οριζόντια ζητήματα. Είναι σημαντικό να δούμε ποιος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος της έρευνας και της ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τη βασική έρευνα βεβαίω, αλλά πρέπει και να επικοινωνήσουμε καλύτερα για τα αποτελέσματα καθώς και να διαδώσουμε τα καλά αποτελέσματα στην κοινωνία. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης να στηριχθούν προγράμματα τα οποία είναι σε πιο αρχική φάση, ε, γιατί είμαστε σε μια φάση ο αναβρασμού σε επιστημονικό επίπεδο, είμαστε ε, ε, και, και μόνο, στην αρχική φάση φαίνονται, διαφαίνονται οι προοπτικές που θα οδηγήσουν ε, σε εμβάθυνση της γνώσης και στην ανταγωνιστικότητα. Πρέπει λοιπόν να αναδούμε και ένα κομμάτι του ρίσκου που θα δώσει αποτελέσματα στο μέλλον. Πρέπει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να διεισδύσουμε σε αυτό το κέλυφος ε, των καινούριων προγραμμάτων ώστε να δούμε τι ορίζοντες διανοίγονται. Επίσης έχουμε έτσι δυνατότητα να συνδυάσουμε εθνικά κονδύλια με τα ευρωπαϊκά και οι κανόνισμοι θα πρέπει να, ε, να ε, τροφοδοτούν αυτές τις ε, ΣΔΙΤ Μάλιστα υπάρχουν εδώ ε, που είναι παραδείγματα αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά οι κανονισμοί πρέπει να είναι κατάλληλοι για να μπορέσουν όντως να εστιάσουν στην προστιθέμενη αξία και να κινητοποιήσουν τις κοινωνίες. Και φυσικά και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μας οδήγησαν να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και να βελτιώσουμε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, κατάλαβα μιλάτε για τα προγράμματα. Το πρίμα, ναι, είναι το project για έρευνα και καινοτομία. Κύριε Ματίας, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την, ε, την ε, Και Εγώ δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην αποστολή αυτή που έγινε στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, παρότι είμαι σκιώδη εισηγήτρια για την αναθεώρηση του ορίζοντα 2020, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, δεν ήμουν εκεί αυτές τις ημερομηνίε της επίσκεψης. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την, τον debriefing που μας έκανε. Και όταν εργαστήκαμε στην προηγούμενη θητεία είχαμε παρόμοια ε, προβλήματα και κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν με εντυπωσιάζει τα όσα είπε. Είναι σημαντικό ωστόσο να έχουμε αυτές τις πληροφορίες γιατί ορισμένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα στη διάρκεια της συζήτησης του ορίζοντας 2020 εξακολουθούν να είναι τα πιο δύσκολα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Για αυτή την ενδιάμεση λοιπόν αναθεώρηση του προγράμματος είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε στο θέμα της διάρθρωσης και της συμπληρωματικότητας ανάμεσα στα διευθυντικά ταμεία και τα ε, κονδύλια τα οποία έχουν ε, αναλυθεί στο πλαίσιο του ορίζοντας 2020, τη φάση της αναθεώρησης των κανονισμών. Τέτοιο είδος σύγχυσης, όπως περιγράφει και εδώ, ε, είναι αυτό που μας δείχνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο η συμπληρωματικότητα δεν θα πρέπει να, να, να, να εννοηθεί ως υποκατάσταση των κονδυλίων. Το θέμα της προσέγγισης είναι επίσης πολύ σημαντικό για την επεξεργασία. γιατί διαφορετικά μπορεί να μην φτάνουν ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που είναι πολύ σημαντικές για τις δύο χώρες μας. Το θέμα της αποκέντρωσης των πόρων επίσης είναι πολύ σημαντικό. Εξακολουθούμε να έχουμε ε, κεντρική μεγάλη πίεση. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε Μιλάμε για διαγωνισμούς, μιλάμε για βοήθεια, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια παραγωγή συστηματική και να μιλάμε μόνο για το ίδιο θεσμούς και τις ίδιες χώρες. Τελευταία μου παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, τελευταία Πρόεδρε, γιατί είναι σημαντική. Είχαμε διάφορες εκθέσεις μέσα στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 και σε αυτή την αναθεώρηση έχουμε μόνο μια έκθεση. Σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κανονισμό υπήρχε ένα αποκλειστικό για τους κανόνες ε, εξέτασης και η συγκήτρια μίλησε για κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει κάτι να αλλάξει εδώ, ε, να αλλάξουν εδώ οι κανόνες συμμετοχής. Δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες συμμετοχής για τις δημόσιους ε, φορείς, όπως τα πανεπιστήμια και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι το ίδιο το σημείο εκκίνησης. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο Ζητώ μάλλον να υπάρξει μια διαβούλευση και να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Γιατί προφανώς δεν λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ladies and gentlemen. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί με την συνεδρίαση των συντονιστών και στις 10 με τις ψηφοφορίες στην Επιτροπή μας στην Ήτρε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν τόσο υπομονετικοί.